Sí, buenas tardes a Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Παρακαλώ να καθίσετε σιγά σιγά. Vamos a Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας της Επιτροπής Αλίας. Λοιπόν, πρώτα έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σας προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με τις εξής τροποποιήσεις. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Καπούλα Σάντος ε, με τη σύμφωνη γνώμη της κυρίας Πρεσδιέ μου ζήτησε διακόπτεται η πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο να τροποποιηθεί η σειρά των σημείων 7 και 8 να αλλάξει η σειρά τους μετά από το σημείο 6 θα περάσουμε αμέσως στο 8 που είναι το θέμα του κυρίου Καπόλας και μετά στη συνέχεια θα δούμε τα τεχνικά μέτρα το 7 το 13ο σε σχέση με τον κύριο Γκάλαγκερ για την χωρίση απαλλαγή του προπολογισμού 2009 για την κοινοτική υπηρεσία ελέγχου της Αλίας θα γίνει μια παρουσίαση από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και όχι από τον κύριο Φώστερ και όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά από έτοιμα διάφορων ευρωβουλευτών της Επιτροπής μας και σύμφωνα με τον εισηγητή, το 13ο θα επισπευστεί στις 9 πριν από το σημείο 11 αύριο στις 9 ε, ναι. και μετά με έτοιμα Φερέιρα σύμφωνα με τις πολιτικές ομάδες θα αναβληθεί για τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου η ψηφοφορία για την πρόταση για τα οικονομικά μέτρα που εισηγητής είναι φυσικά ο κύριος Φερέιρα. Ναι κύριε Ρωμέβα παρακαλώ συσχετίζεται με την ημερήσια διάταξη της αύριο. Είναι ένα μικρό αίτημα που έχω, διότι στο 11 έχουμε τη συζήτηση της γνωμοδότησης για τη συμφωνία, τη συμφωνίας με το Μαρόκο, στο, συγγνώμη, στο 12, για τα αμοιβαία μέτρα για τα γεωργικά προϊόντα. Ξέρω ότι υπάρχει νομοθετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με συμφωνία Λίας που ε, συνάπτεται με αυτό. Το αίτημά μου θα ήταν λοιπόν αυτό αύριο κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πληροφορήσουν για τη νομική γνωμοδότηση που έχουν σε σχέση με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Αυτό το αίτημα είχα απλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαρίστω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πληροφορήσει και να ενημερώσει για το θέμα εσείς, ε, που είσαστε εσείς εισηγητής. Δεν έχει καμιά σχέση όμως με τη Συμφωνία Αλίας δεν έχει κάποια σχέση, αλλά τέλος πάντων, αφού αυτό είναι το έτοιμά σας, οποιαδήποτε πληροφόρηση σε σχέση με αυτό θα είναι ενδιαφέρουσα για τα άλλα μέλη. Θα δούμε. Λοιπόν, με αυτό εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και περνάμε έτσι λοιπόν στη συνέχεια στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 26ης-27ης Οκτωβρίου και 8ης-9ης Νοεμβρίου. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασής μας δεν υπάρξει καμιά αντίρρηση, καμιά ένσταση, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται. Στη συνέχεια έχουμε τι ανακοινώσει τη Προέδρου. Δεν έχω καμιά ανακοίνωση να κάνω. Και έτσι περνάμε αμέσω στο σημείο 4 της ημέρησια διάταξης, που είναι η έκθεση του κυρίου Γκάλαγκερ για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής που προβλέπεται να ψηφιστεί σήμερα. Κάποιες τοπολογίες σε σχέση με την έκθεση Γκάλαγκερ Δίνω τον ε, λόγο στον κύριο Γκάλαγκερ για να περάσουμε στην ψηφοφορία στη συνέχεια. Ελπίζω ότι όλοι θυμηθήκατε να φέρετε τις κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κύριε Γκάλαγκερ, έχετε τον λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση αντιμετώπισε πάρα πολλές αντιφατικά σχόλια επειδή των προφοριών που προέρχονται από τον τομέα και ίσως και εσείς ε, να είστε σε θέση, κυρία Πρόεδρε, σήμερα να μας δώσετε μια περιγραφή ή να μας ενημερώσετε για τις τελευταίες προφορίες που είχατε στην ε, συνάντηση με τις χώρες ΑΚΕ. Αυτό είναι υπάρχει μόνο το ένα σχόλιο. Και δεύτερο, από ό,τι καταλαβαίνω η λόγω συμφωνία δεν έχει υπογραφεί ακόμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Φιλής και κατά συνέπεια το, Συμ... το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να ζητά την συνένεση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 2.18 κάθος 6, ούτε υπάρχει κάποια ένδειξη αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μήπως θα μπορούσε λοιπόν κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφινιστεί εάν έχει υπογραφεί ή όχι. Εάν δεν έχει υπογραφεί είμαστε, ε, έχουμε κάποια υποχρέωση να εγκρίνουμε τη συμφωνία αυτή. Από όσα γνωρίζω για το θέμα είναι τα εξή. Σε σχέση με την εφαρμογή της διαδικασίας σε σύμφωνης γνώμη στο Συμβούλιο, δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση για να προσυπογράψει μια συμφωνία. Όταν θα έχει δοθεί αυτή η συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπογράψει ή δεν θα υπογράψει. Αλλά καταρχήν πρόκειται για το θέμα υπογραφής μιας συμφωνίας εδώ. Και εμείς εμείς δεν θα μπορούσαμε, όπως έγινε σε σχέση με τις νήσους Σολομώντα, να περάσει η έκθεση στην Ολομέλεια. Μπορεί να ψηφιστεί σήμερα, δεν θα μπορούσε όμως να περάσει στην Ολομέλεια μέχρι ότου το Συμβούλιο από πλευράς του θα το ζητήσει ως αίτημα επίσημα από μας να γίνει. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προσυπογράψει συμφωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Χιλή και στη συνέχεια θα πρέπει το Συμβούλιο να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να υπάρξει ε, η διαδικασία σύμφωνη γνώμη. Αυτό δεν παρακολεί σήμερα να μπορέσουμε να ψηφίσουμε και να επισπευστεί αυτό το θέμα από πλευρά Ευρωπαϊκής, από Επιτροπής. Το μόνο είναι που δεν μπορεί να περάσει στην Ολομέλεια μέχρι ότου ζητηθεί αυτό από το Συμβούλιο. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση, θα περάσουμε τώρα στην ψήφιση αυτή τη έκθεση. Εντάξει. Και θα δούμε θα ζητήσει, αν θα ζητήσει το Συμβούλιο να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη. Και έτσι θα περνούσαμε στην Ολομέλεια, την αντίστοιχη Ολομέλεια του Δεκεμβρίου ή του Ιανουαρίου 2011. Θα το δούμε αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γιατί δεν εξαρτάται από εμά αυτό. Από μένα δεν εξαρτάται. Λοιπόν, αν συμφωνείτε κύριε Γκάλαχερ, να ψηφίσουμε τώρα στη συνέχεια να διευθετηθεί αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε μια τροπολογία, την υπαριθμόν 1, <clears throat> όσον αφορά την παράγραφο 1 Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν επ' αυτής. Α, συγγνώμη κύριε Γκάλαχερ, συγγνώμη. Okay, κύριε Πρόεδρε, ε, ναι, αποσαφηνίστηκε το θέμα. Αλλά ας δούμε λίγο και τις εναλλακτικέ. Εάν εγκριθεί σήμερα από την Επιτροπή μας και υπογραφή από το Συμβούλιο η συμφωνία αυτή με τη Χιλή, εάν την απορρίπτουμε όμως σήμερα, τι συμβαίνει. Μπορεί η Χιλή και το Συμβούλιο ερήμηνη μόνο να συνεχίσει και να προχωρήσει η υπογραφή. Γιατί πραγματικά αυτό είναι εμπεγμός του να λάβουμε τώρα μια απόφαση. Ξαναγυρίζουμε δηλαδή στα πρώτη συνθήκη. Λοιπόν, προσέξτε, θα σας το εξηγήσω. Αν υποθέσουμε ότι ψηφίζουμε σήμερα και απορρίπτουμε αυτή την πρόταση, υπό αυτή την υπόθεση, γιατί αν εγκριθεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υποθέτοντας ότι απορρίπτεται λοιπόν σήμερα η πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα και έτσι μπορεί να προσυπογράψει και θα ξεκινούσε η συμφωνία να εφαρμόζεται προσωρινά, με προσωρινό χαρακτήρα. Μέχρι ότου το Κοινοβούλιο θα έχει τελικά γνωμοδοτήσει δίνοντα σύμφωνη γνώμη από πλευρά του. Στην οποία περίπτωση, αν αποφασίσει όχι το Κοινοβούλιο, φυσικά αυτή δεν θα, δεν θα αρχίσει να ισχύει η συμφωνία. Αν γνωμοδοτήσει όχι το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι πιστεύω. Ότι αν, αν τώρα πει όχι το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, αν πει όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα οδηγούσε αυτό το θέμα στην σε υπογραφή. Αυτή είναι όμως η προσωπική μου άποψη σε σχέση με την εκτίμηση του τι θα μπορούσε να συμβεί. Okay. Λοιπόν, εντάξει, πολύ καλά. Για να δούμε. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Λίγη ψηφοφορία. Τι συνέβη με τις οθόνες. Λοιπόν, για άλλη μια φορά άρχεται η ψηφοφορία. Επαναλαμβάνουμε. Κάτι συνέβη εδώ με τις συσκευές. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 14, 5 υπέρ, 14 εναντίον, μια εποχή Γι' αυτό ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο ψηφίσματος, σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος του εισηγητή. Παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εδώ εγκρίνεται 15 ψήφοι υπέρ, 5 εναντίον. Συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή Αλίας απέρριψε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Χιλή. Ευχαριστώ. Και αυτό θα διαβιβαστεί στην αντίστοιχη ολομέλεια όταν θα η ώρα. Λοιπόν, για τον Ιανουάριο προβλέπετε, αλλά σας λέω ότι πρέπει να αναμείνουμε να δούμε το αίτημα επίσημα του Συμβουλίου, πότε θα διατυπωθεί. Και έτσι ολοκληρώνεται, ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες για σήμερα. Και περνάμε στο σημείο 5 τη σημερινή διάταξης. Ησυχία λίγο παρακαλώ, εντάξει. Περνάμε στο σημείο 5, έλεγα, της ημερήσιας διάταξης που αναβλήθηκε. Και έτσι περνάμε στο σημείο... Παρακαλώ λίγη ησυχία. Περνάμε στο 6 της ημερήσιας. Μα τι γίνεται. Τώρα δεν είναι ο Γαρίγα Πογέδο, λέει εδώ. Eh, λοιπόν, εντάξει απίθανο και απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με την Επιτροπή Αλίας. Στο 6 είναι σε συνάντηση συντονιστών ο κύριος Γκαρίγα Πολιέδο. Δεν μπορεί να προσέθει αυτή τη στιγμή. Αναβάλουμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Ο κύριος Γκαρίγα που είχε πει θα ερχόταν δεν μπορεί να προσέθει τώρα. Περνάμε στο σημείο 8 τώρα της ημερησίας διάταξης που είναι η έκθεση του κύριου Καπούλα Σάντος για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ένωσης των Κομορών. Κομορών Νήσων. <clears throat> Στην πρόταση τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την παρουσίαση... Α, όχι. Τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτή, να σας εξηγήσω εγώ τι γίνεται, θα το αναβάλουμε το σημείο κακ αυτό της ημερήσια διάταξης. για την πληροφόρηση τι συμβαίνει με την ΙΚΑΚ. Τι θέλετε να κάνουμε, δεν φταίω εγώ. Έτσι είναι το θέμα με την αλία. Να συζητηθεί, να αναφερθεί το τι συνέβη με την ΙΚΑΚΑ. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε λοιπόν, υπήρξε μια συνεδρίαση της ΙΚΑΚΑ με την... Ε, ε, είναι έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει. Πραγματικά το λέω προσωπικά. Εγώ είμαι υπέρ της αλληλείας εδώ. Είναι πραγματικά όνειδος αυτό. Εγώ ως πρόεδρος παραπονούμε εδώ για όσους δεν ενδιαφέρονται και δεν παρακολουθούν. Αν δεν παρακολουθούν και δεν ενδιαφέρονται Λοιπόν, σας έλεγα ότι η συνεδρίαση της ΙΚΑΚΑ, Περιφερειακή Οργάνωσης Αλίας, που ασχολείται με τα αναστευτικά είδη του Ατλαντικού και της Μεσογείου, που συνήθιε την προηγούμενη εβδομάδα, 26-27 Νοεμβρίου, στο Παρίσι. Είχε την ετήσια συνάντησή της και είχαμε μια αντιπροσωπεία αρκετά πολύ άριθμη και ο κύριος Σάντσιος Πρεσέντο, ο κύριος Καντέκα, Αρσένη, ο κύριος Ρωμέβα, εγώ η ίδια, συμμετείχαμε και να σας πω σχετικά ότι εμείς πιο πριν από αυτή τη συνεδρίαση είχαμε ζητήσει μετά από τα προβλήματα που γνωρίζετε ότι υπήρχαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για την τελική εντολή που είχε δοθεί από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μας είχε αρνηθεί την εντολή και γνωρίζαμε ότι είχε υπάρξει μια απόρριψη σε σχέση με το σχέδιο εντολής που είχε υποβληθεί από την Επίτροπο Δαμανάκη. Θέλαμε παρόλα αυτά να έχουμε την τελική εντολή του Συμβουλίου στα χέρια μας, αλλά δεν ήταν δυνατόν αυτό λόγω των διοργανικών σχέσεων που διαρκώς μετά από την έναρξη σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας βλέπουμε σε αυτό το κοινοβούλιο στι σχέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου. Μετά από αυτά θα σα πω ποιε ήταν οι πρώτες οι αποφάσεις οι πιο σημαντικές που ελήφθησαν μέσα στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης και όπως υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που είχαν συμμετάσχει μπορούν να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν τις απόψεις μου, τα όσα θα σας πω αν χρειάζεται. Πρώτα απ' όλα με το αστέρι για όλους που ήταν ο ερυθρόπτερος τόνος της Μεσογείου, του Ατλαντικού, Ανατολικού Ατλαντικού και όπως όλοι γνωρίζετε σχετικά το ΤΑΚ που υπήρχε για εφέτος ε, για συγκεκριμένο όγκο ε, τόνων ε, με την έγκριση μια σύσταση που είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος συμφωνήθηκε να είναι 12.900 τόνοι. Αυτοί οι 12.900 τόνοι στο τέλος τέλος ήταν λιγότεροι γιατί υπάρχουν συμβαλόμενα μέρη τα οποία απεσύρθησαν και είπαν δεν θα εξαντλήσουν την ποσοστοσή τους. Επιπλέον υπάρχουν και κάποιες επιστροφές από κάποιες χώρες ε, για τη Γαλλία, Ιταλία, για να μην αναφέρω άλλους που πρέπει να επιστρέψουν μέρος των ποσοστώσεών τους ε, και γι' αυτό η δυνατότητα να επιτευχθεί ο στόχος της βιομάζας της μέγιστης ε, απόδοσης, αηφόρου απόδοσης με ένα 60% ίσως και θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια αύξηση μια και στο τέλος ε, το τελικό τάκ θα είναι μικρότερο από αυτό που εγκρίθηκε. Επιπλέον για να ε, κατοχυρώσουμε, να εγγυηθούμε την υλοποίηση τα συμβαλόμενα μέτρα θα πρέπει να υποβάλουν ένα ετήσιο πρόγραμμα αλληλεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και την και σε περίπτωση που απορριφθεί αυτό το πρόγραμμα γιατί δεν θα συμμορφώνεται σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές με τους στόλους ε, θα, από πλευράς στόλων θα υπάρξουν αυτές οι προσαρμογές. Έτσι λοιπόν έχουμε την κλίδα κατανομής ε, ε, για την ΤΑΚΑ που δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλγερία μόνο μείωσε το ποσοστό της, μειώθηκε και για την ε, Λιβύη, Μαρόκο και Τουρκία έχει αυξηθεί. Σε σχέση με τα μέτρα ελέγχου που προτείνονται και εγκρίνονται, είναι πολύ πιο αυστηρά από εκείνα τα οποία υπήρχαν και ίσιαν μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, σήμερα η κάλυψη με επόπτε ε, που θα διασφαλίζεται για να ε, καλύπτονται και τα ρημουλκά, καθώ επίση και η κάλυψη με του επόπτε που θα ασχολείται με τα παραγαδιάρικα επίσης. Και αυτές είναι οι κυριότερα μέτρα που υιοθετήθηκαν γύρω από αυτό που είναι το θέμα του ερυθρόπτερου τόνου. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι το θέμα του, της, των αλευμάτων στον κόλπο της ε, Γουινέας. Είχαμε και την, ε, ε, τις δράσεις στα διαβήματα της Ευρωπαϊκής, Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του... της Ιαπωνίας. Φαίνεται ότι σε αυτή τη ζώνη του Ατλαντικού υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα της ε, αλίευσης και μεταφοράς από τον Ινδικό ωκεανό στον Ατλαντικό με τα προβλήματα που υπάρχουν ε, λόγω της πειρατείας ε, στον Ινδικό. Έχουν μετατεθεί λοιπόν στον Ατλαντικό. Υπάρχει αύξηση του δυναμικού, κυρίως της Κίνας σε αυτά τα ύδατα αύξηση του δυναμικού. Υπάρχει σημαντική ε, σύλληψη αλληλεία γόνων ψαριών έλλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις και υπεραλίευση λόγω έλλειψης σεβασμού των κανόνων. Και βλέπουμε ότι αυτοί που αλλιεύουν εκεί έχουν δηλώσει συμβαλόμενα μέρη πάνω από 110 αύξηση της αλίευσης. Έχουν δηλαδή ένα, ε, μια ποσόστοση 5.000 τόνων και δηλώθηκε ότι πάνω από 10.000 τόνους αλλιεύουν. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία πρότειναν μια σύσταση που εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα όπου εξετάζεται μια νέα ζώνη απαγόρευσης αλλιείας νέα ζώνη απαγόρευσης κυρίως για να αποφύγουμε την αλίευση γόνων ε, νέων ψαριών, ε, μικρών ψαριών και έτσι θα πρέπει να προστατευτεί η παραγωγή γόνων και να διασφαλίζεται αυτό και με την παρουσία εποπτών. Αυτό απορρίφθηκε από μέρος των συμβαλωμένων μερών και από τις Ηνωμένε Πολιτείες που όπως ξέρετε έχουν σημαντικά συμφέροντα με την Γάνα, εμπορικά συμφέροντα και έτσι απερίφθη από αυτού ε, τα μέτρα ελέγχου τα οποία είναι απαραίτητα όμω, ώστε να συμμορφώνονται τα να συμμορφώνεται η αλλιευτική δράση. Γι' αυτό απέσυραν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία την πρότασή του μια και δεν υπήρχε απαρτία και έτσι εγκρίθηκε μια παράταση ενός έτους ε, ακόμα της σημερινής κατάστασης των πραγμάτων του status quo. Είναι θλιβερό αυτό για την κατάσταση των αλλιευμάτων σε αυτήν την περιοχή. Και όσον αφορά την Μεσόγειο υπήρξε πάλι παράταση της σημερινής κατάστασης των πραγμάτων. Θα ήθελα να σας πω ότι το θέμα του ξηφία στην Μεσόγειο, που είναι και αυτό ευαίσθητο θέμα, είναι όνειδος ότι δεν ελήφθη καμία απόφαση σχετικά. Και σε σχέση με τις ωκεάνιες ζώνες ανακοινώθηκε ούτως ή άλλως αυτό, αλλά έχω εδώ και μία πληροφορία για τον ερυθρόπτερο ε, τόνο σχετικά Όσον λοιπόν αφορά τον ξηφία στην, στον Βόρειο Ατλαντικό, πάλι δεν ελήφθη καμία απόφαση, παρότι εφέτος έπρεπε να είχε διεξαχθεί μια κατανομή, μια νέα κατανομή των μια νέα, ένας νέος επιμερισμός ποσοστώσεων και επίσης υπήρξε ένα roll over όπως λένε, μια παράταση δηλαδή της σημερινής κατάστασης των πραγμάτων. Και το θέμα των καρχαριών είναι ένα θέμα που απασχόλησε είναι τα αστέρια βλέπετε της παράστασης οι καρχαρίες και οι αποφάσεις είναι οι εξή Το Μαρόκο και που είναι ένα από τα ε, αφορά τα αλλιεύματα αυτά ζητήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή να συντάξει μια αξιολόγηση ε, αυτών των αποθεμάτων και να υπάρξει μια παρακολούθηση των επιπέδων αλληλείας, ετήσιων επιπέδων αλληλείας που θα ε, δίνουν τη δυνατότητα της μέγιστης ε, αηφορίας όσον αφορά τα ετήσια αλλιεύματα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζουν να λαμβάνονται μέτρα από το Μαρόκο και σε σχέση και με πληροφορίες που υπάρχουν ώστε η Επιστημονική Επιτροπή να μπορεί να αξιολογήσει αυτό το αλίευμα για το άμεσο μέλλον. Όσον αφορά τον ωκεάνιο Καρχαρία, όσον αφορά την ε, εμπορία του υπήρξε μια συμφωνία για τον ε, Καρχαρία, το σφυροκέφαλο ε, Καρχαρία για την, μια κάποια ελαστικοποίηση για τα συμβαλόμενα μέρη όσον αφορά τα παράκτια κράτη τα οποία βρίσκονται υπό ανάπτυξη, είναι αναπτυσσόμενα κράτη. Αντιθέτως όμως δεν εγκρίθηκε μια πρόταση που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Καρχαρία Αλεπού όπως τον αποκαλούν. Ε, έχουμε και την Περιφερειακή Οργάνωση Αλίας ε, του Ινδικού που απαγορεύτηκε η ε, ε του καρχαρία αυτού εκεί. Ωστόσο όμως σε σχέση με το σφυροκέφαλο είναι διαφορετική κατάσταση. Επίσης μια έγκριση της, μια σύσταση για τις χελώνες και θέματα τα οποία αφορούν εδώ την ε, χελώνα, όχι τον ε, Καρχαρία. Σε σχέση με τις προηγούμενες αναφορές που έγιναν, έγιναν ολοκλήρωσε. έτσι. Θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Συμμόρφωσης για άλλη μια φορά αναφέρθηκαν τα προβλήματα της συμμόρφωσης με τα μέτρα αλίας σε αυτή τη ζώνη και σε σχέση με άλλα συμβαλόμενα μέρη από τα 48 δύο υλοποίησαν. 23 πήρανε μια επιστολή ταυτοποίησης των, κακο, των κακοσκημένων, των προβλημάτων και άλλοι πήρανε μια κάρτα με συστάσεις. Το, για το μεγαλύτερο μέρος αυτών των συμβαλωμένων μερών τα, πράγματα δεν βαίνουν καλώς, βλέπετε, δεν συμμορφώνονται. Και υπήρξε η δυνατότητα σχεδιασμού, πρόταση σχεδιασμού ενός πλαισίου κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αυτά για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την υλοποίηση και τη συμμόρφωση που δεν είναι τέλεια. Και τέλος να σας ανακοινώσω επίσης ότι στο θέμα της ε, ε, έρευνας όσον αφορά τον ερυθρόπτερο τόνο, αλλά υπάρχουν και άλλα προγράμματα ε, υποεξέλιξη για άλλα είδη, αλλιευτικά είδη αλλά για τον ερυθρόπτερο τόνο ζητήθηκαν κονδύλια ώστε να μπορούν με αυτά τα κονδύλια να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα κυρίως ε, όσον αφορά την προοπτική και την έρευνα για τον ερυθρόπτερο τόνο για το μέλλον. Αυτά σε σχέση και με τα προβλήματα που γνωρίζουμε ότι υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησης θεμάτων που αφορούν την αλληλεία ελπίζουμε βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει την δυνατότητα να διατεθούν αυτά τα κονδύλια ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα θέματα για τον ερυθρότερο τόνο, τα προγράμματα αυτά θα μπορέσουν να συνεχιστούν στο μέλλον και αυτές οι έρευνες. Τούτων λεχθέντων τώρα θα έλεγα ότι με αυτά πιστεύω ότι κάλυψα αυτά τα οποία με σύντομη ενημέρωση έπρεπε να αναφέρω στις ανακοινώσεις Προέδρου αν ενδιαφέρεστε για κάποιο θέμα συγκεκριμένα μπορώ να σας ε, το εξηγήσω πιο καταλεπτός ε, ή και να ε, διατεθεί και κάποιο άλλο στοιχείο σε εσά. Είμαι στη διάθεσή σας πάντα για να μπορέσω να σας πληροφορήσω πιο καταλεπτός, πιο εξειδικευμένα. Αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή την επιτροπή μας χρειάζεται αυτό. Εσείς έχετε τον λόγο, το ζητήσατε κύριε Ρωμέβα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Να προσπαθήσω να συμπληρώσω κάποια στοιχεία μόνο και κάποια άλλα να τα σκιαγραφίσω. Ξεκινώντας με ένα πρώτο προβληματισμό γενικά όσον αφορά την ίδια τη δυναμική της ΣΥΚΑΚ. Αυτή είναι η τρίτη συνεδρίαση που είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω και διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ουσίας όσον αφορά τους ίδιους τους κανόνες. Η εντύπωση που αποκόμισα από το θέμα της Επιτροπής ε, Εφαρμογής και Συμμόρφωσης είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το νομοθετικό, το εκτελεστικό και το δικαστικό είναι το ίδιο άτομο ο ίδιο φορέας, το ίδιο σώμα. Και έτσι είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν καλά τα πράγματα. Όταν συντάσσονται οι κανόνες από εκείνον που τους εφαρμόζει και από εκείνον που τους ε, εκδικάζει ή που πρέπει να τους ε, ε, κρίνει ή να επιβάλλει κυρώσεις, έχουμε πρόβλημα. Αυτή είναι η να επιβαλλει κυρώσει, εχουμε προβλημα αυτη ειναι η εντυπωση που έχω σε σχέση με την ΙΚΑΚΑ. Κάπως αυτό συμβαίνει εκεί. Με αποτέλεσμα στο τέλο, στην Επιτροπή εφαρμογή να γίνεται πολύ θόρυβος αλλά να μην υπάρχει πολλή ουσία, να μην βγαίνει ζουμί. <laughs> Υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά όταν προσπαθεί κανείς ε, να καταλήξει κυρώσεις και να τιμωρήσει ε, τα κακό κείμενα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα είδος κάποια συμφωνίας και τα πράγματα δεν πάνε πέρα από διακηρύξεις ε, στο επίπεδο διακηρύξεων. Δεν ακολουθούν πράξεις. Αυτό το θέμα με ανησυχεί και θα έπρεπε να μας προβληματίσει και εμάς θα έλεγα. Όσο αφορά την ουσία, Πραγματικά συμφωνώ ότι τα σημαντικά θέματα ήταν αυτά. Οι καρχαρίες πρώτον, εντάξει, αλλά ε, σε σχέση με τα καλά μαντάτα της συνεδρίασης, τα καλά μαντάτα ήταν ότι τουλάχιστον ένα μέρος ε, των καρχαριών προστατεύονται πλέον. Έγινε δουλειά και από κάποιες οργανώσεις μη κυβερνητικές, μεταξύ αυτών και της ΟΣΕΑΝΑ, ώστε το θέμα να τεθεί στο τραπέζι και να εξεταστεί. Διαπιστώνω μια αντίφαση εδώ. Η πρόεδρος το είπε και η ίδια πιο πριν στο ότι έχουμε ένα είδος προστατευμένο, καλύτερα προστατευόμενο, Αντίθετα όμως έχουμε άλλα είδη τα οποία δεν ε, την χάνουν αυτής της ε, προστασίας. Υπάρχει κάποια συμβατότητα, κάποια ασυνέπεια και πρέπει να βελτιώσουμε αυτά τα πράγματα. Πέρα από τις θλιβερές ε, εξαιρέσεις όπως τον Αλεπού Καρχαρία Αλέπου. Είναι όμω αυτή η καλή είδηση, τα καλά μαντάτα από την ΙΚΑΤ στο Παρίσι. Όσον αφορά τον Ξηφία, συμπίπτει η άποψή μου με τη Προέδρου. Όσον αφορά την κατάσταση που είναι πολύ σοβαρή, όπως και του ερυθρόπτερου ε, τόνου στη Μεσόγειο, είναι θλιβερό γιατί δεν εγκρίθηκε τίποτα. Και αρκετέ οργανώσει είχαν ζητήσει να εγκριθεί κάτι. Και είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε ότι το χρονόμετρο, το ρολόι συνεχίζει να μετρά τον χρόνο, πιέζει ο χρόνος, προχωρεί ο χρόνος ε, και δεν γίνεται τίποτα και για κάποιε ίδιε πρωτοβουλίε του ιδίου του τομέα από πλευρά τη ευρωπαϊκού τομέα που δεν έγιναν δεκτέ από του άλλου τομεί, ε, από ε, του ομολόγου του. Αυτό είναι λοιπόν κάτι σωστό και πρέπει να το επισημάνουμε. Και για το τελευταίο, ερυθρόπτερο τόνο. Για μένα εδώ υπάρχουν τρία σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι η αναθεώρηση των ποσοστώσεων. 12.900 ε, τόνοι ε, και όσον αφορά αυτό πραγματικά λαμβάνοντας υπόψη ε, τις, το, τις πιθανότητες που πρέπει να εξετάσουμε δεν υπάρχουν πώς θα εξετάσουμε την πιθανότητα να γίνει κάτι ή όχι για έναν τομέα. Πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει, είναι αναγκαίο νομίζω αυτό, να συνειδητοποιήσουμε τα επίπεδα πιθανοτήτων ε, που ε, οδηγούν σε υπολογισμούς ε, και καταλήγουμε σε χαμηλά επίπεδα. Να κάνουμε την ερώτηση, αν εμείς είχαμε 60% μπαίναμε σε ένα αεροπλάνο που μόνο 60% πιθανότητες θα είχε να έφτανε στον προορισμό του, δεν θα μπαίναμε σε αυτό. Πρέπει να αξιολογηθεί λοιπόν στο βαθμό στον οποίο μπορούν τα πράγματα να πάνε καλά ή όχι. Και μένω και επιμένω για το καλό, το καλό το να έχει υιοθετηθεί ένα ποσοστό 6.000 και κάτω. Δεν υιοθετήθηκε αυτό και δεν μπορώ να το θεωρήσω θετικό. Το δεύτερο και είναι θετικό είναι το payback και σε σχέση και με τη Γαλλία εδώ πραγματικά ε, διαφορώ, έχω διαφορετική άποψη με κάποιους Γάλλους συναδέλφους αλλά παρόλα αυτά, παρόλα αυτά είναι ένα καλό μαντάτο ότι δεν, ε, ε, δεν συγχωρήθηκε αυτό το payback γιατί θα ήταν κακό προηγούμενο θα ήταν κακό προηγούμενο. Αν σε μια κατάσταση όπου είναι περίπλοκο το πράγμα, αρχίζουμε να συγχωρούμε, να διαγράφουμε τα χρέη και να ξεχνάμε το τι πρέπει να γίνει. Δεν είναι καλό λοιπόν. Και για τον ε, τόνο λοιπόν ε, είναι καλό το ότι δεν συγχωρέθηκε το payback, ε, δεν συγχωρέθηκε, δεν διαγράφηκε το payback στη Γαλλία δεν είναι μόνο το θέμα της Γαλλίας, είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είχε κατανεμηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το είχε πάρει η Γαλλία. Και εδώ τώρα ως υποσημείωση κάτι θα ήθελα να πω, είναι το θέμα των ε, προστατευόμενων ζωνών και των απαγορευμένων περιοχών. Είχε τεθεί κάποτε στο παρελθόν, είναι ένα θέμα ενδιαφέρον, σημαντικό, αναγκαίο. Στη συνεδρίαση απλά αναφέρθηκε η ανάγκη να μελετηθεί η κατάσταση, λέει, αν, να δούμε αν σε ένα μέλλον ε, απότερο μέλλον θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη αυτό το μέτρο. Εγώ εμένω και επιμένω αυτό το θέμα θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον και θα πρέπει στο μέλλον να μην το αγνοήσουμε, μην το ε, διαγράψουμε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ευχαριστώ. Merci, ε, Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι συμμετείχα και εγώ σε εκείνη την επιτροπή ε, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Δυστυχώς πάρα πολλές αποφάσεις αναβλήθηκαν για του χρόνου σε πάρα, πολλές, πάρα, πολλές, πάρα πολλά θέματα. Σε αυτό που είπατε, κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ. Δηλαδή υπάρχει μια πτώση ε, σε ό,τι αφορά τα λεύματα ξυφιών για τα οποία δεν είχα ληφθεί αποφάσεις. Αντίθετα, και εδώ συμφωνώ με τον προαλήσαντα συνάδελφο, Μα συμβαίνει να συμφωνούμε από και καιρό τέλο πάντων ότι η ποσόσταση των 12.900 τόνων, εάν το συγκρίνουμε με τους 13.500 τόνους που είχαν γίνει αποδεκτοί πέρσι και που σας, ε, υποδι... σας ε, ε, είχα λάβει ήδη υπόψη μια μείωση κατά 40% των αλλιευμάτων, είναι μια ποσόσταση που κατά απόλυτα λογική και επομένως αποδεκτή από τους πάντες. Αντιθέτως, προφανώς σε ό,τι αφορά τις ε, ε κάτω χώρες, ο Ραούλ, όπως είπε πολύ σωστά, η εξάλληψη των χρεών δεν είναι δεν είναι ουσιαστικά εξάλληψη διαγραφή χρεών, είναι διαφορετική, διαφορετική κατανομή των αποπληρωμών. Θα μπορούσε να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια κλιμάκωση σε μια τετραετία της ε, καταβολής ε, ε, των, και επιστροφής των φόρων αυτών, που θα επέτρεπε βέβαια την επιβίωση κάποιες από τις χώρες αυτές, γιατί είναι πολύ μεγάλο οικονομικό, χρηματοοικονομικό και κοινωνικό σοκ το οποίο επιφέρεται και είναι πραγματικά δραματικό για την γαλλική ελία, γενικά του γαλλικού τόνου. Υπάρχει λοιπόν, αν θέλετε, ένα αντιφατικό και μετριασμένο συνέστημα ε, ικανοποίηση σε ό,τι αφορά την ποσόσταση και απογοήτευση στο ότι δεν υπάρχει μια κλιμάκωση των χρεών. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για διαγραφή χρέου αυτό που ζητάμε, αλλά μια κλιμάκωση των αποπληρωμών. Πέραν όλων αυτών, η όλη συνάντηση με την ε, συμφωνία, την ε, Γενική Συμφωνία ΓΚΑΤ, έλαβε χώρα και σε πολύ καλό πνεύμα. Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Εντάξει. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτό το θέμα και κυρίως επειδή είχα υποσχεθεί στον κύριο Καπόλος ότι πριν από τις 4 θα εξετάζαμε το δικό του θέμα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να κάνουμε λόγο για την ΙΚΑΤ αν επιθυμείτε, εντάξει. Bueno, si no, eh? Δεν είναι εδώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν δεν παρίσταται δεν μπορούμε να έχουμε την παρουσίαση του πρωτοκόλου. Α, εσύ είσαι μεσία Μίλατ. Μάλιστα, κύριος Μίλατ. <laughs> On a parlé du Mais non, mais ce n'est pas pour que δεν ήσασταν εδώ δεν θα ήσασταν για την συμφωνία 4, δεν είναι, θα ήσταν για τις Κομόρες. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα υπάρχει κάτι. Αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. να καθίσει. Ναι, πρόεδρος. Δεν μπορούμε έτσι να τα μεταχειριζόμαστε τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί όχι, ρωτάω παρακαθημένος. Eh, λοιπόν, περνάμε λοιπόν στο 8 της ημερήσιας διάταξης. Το πρωτόκολλο για να συνεχιστούν οι δραστηριότητες αλλίας με την, τα αντισταθμίσματα τα οικονομικά όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ίσων Κομορών. Όπως ξέρετε αυτό το πρωτόκολλο είχε αναδιαπραγματευτεί και δίνω τώρα από πλευρά τη Σοσιαλιστικής Ομάδας ο εισηγητής είναι ο κ. Καπόλας θα πάρει τον λόγο ο κύριος για να παρουσιάσει την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με αυτό το πρωτόκολλο. Έχετε, μητάτε τον λόγο και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Αλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πάντοτε χαρά για μένα να πάει βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Ελίας ε, και είμαι στη διαθεσία σας ε, πάντοτε και οποιαδήποτε ώρα μου πείτε να έρθω σχετικά με το θέμα αυτό, με αυτήν την Συμφωνία Ηλίας με τις Κομόρες, με την Ένωση των Κομορών. Αυτό βεβαίως είναι σε μια αλληλευτική ζώνη, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για τον Ευρωπαϊκό Στόλο, εφόσον υπάρχει μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών πλοίων ε, που δραστηριοποιούνται στον Ινδικό Ωκεανό ε, κυρίως ε, που αλλιεύουν ευθύνοειδή σε μια περιοχή που σήμερα διαταράσσεται από την πειρατεία και η οποία σχετικά με την πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα εξαρτάται από την Indian Ocean Tuna Commission, την Επιτροπή ε, Θηνοειδών για τον Ινδικό Ωκεανό. Αυτό το νέο πρωτόκολλο με τις κομόρες είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο θα, έχει, θα έπρεπε να έχει μια διάρκεια τριετή οι ε, δυνατότητες οι αλλιευτικές έχουν σχετικά μειωθεί σε σχέση με τις προηγούμενες δυνατότητες εφόσον για να ε, υπολογίσουμε ε, την αξία ήταν 6.000 τόνοι ενώ τώρα έχουμε 4.800 τόνους πράγμα που αντικατοπτρίζει την δραστηριότητα στην προηγούμενη περίοδο των πλοίων μας, των σκαφών μας. Ο αριθμός όμως των πλοίων που έχουν άδεια να αλλιεύουν έχει αυξηθεί και πέρασε από 58 σε 70 πλοία από 40 ε, για παραγάδια ε, και ε, τα υπόλοιπα είναι ναυύρια γρήπων η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συμφωνία αυτή ε, δεν θα μειωθεί, θα περάσει σε 615.000 κατέτος, 315.000 για την πρόσβαση στις πηγές και 300.000 για την υποστήριξη στην πολιτική ε, της αλληλείας Υποστηρίζουμε λοιπόν τις προσπάθειες αυτές. Υπάρχει επίσης μια αύξηση των συνεισφορών, των τελών που πληρώνουν οι εφοπλιστές για την δραστηριότητά τους στην περιοχή. Τα νέα στοιχεία στο πρωτόκολλο αυτό σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο είναι τα εξής. Έχουμε μια ρήτρα αποκλειστικότητας που εισήχθη Δηλαδή δεν είναι δυνατόν για, τους, για τα ευρωπαϊκά πλοία να αλλιεύουν άλλα είδη από αυτά που προβλέπονται ε, στο, στη συμφωνία, δηλαδή τον τόνο. Υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρησης της συμφωνίας που εισήχθη για την περίπτωση ε, σημαντικής αλλαγής στην πολιτική της αλίας, ούτως ώστε να μπορούμε ανα πάσα στιγμή ε, να αναθεωρήσουμε το πρωτόκολλο αν ε, έχουμε μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και επίσης μια ρήτρα αναστολής ε, καταγγελίας ε, της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις ε, διατάξεις της συμφωνίας της Κοτονού και τις διατάξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη συμφωνία της Κοτονού. Επίσης υπάρχει μια ρήτρα αναστολής, διακοπής της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση μη τήρησης των προηγουμένων διευθετήσεων ως προς την υποστήριξη της πολιτικής και των στόχων της αλλιευτικής πολιτικής που προσπαθούμε να υποστήριξουμε μαζί με τη χώρα αυτή. Άλλο στοιχείο που πρέπει να επισημάνω θα υπάρξει σε κάθε πλοίο που θα δραστηριοποιείται στη ζώνη αυτή ένας ναυτικός από τις Κομόρες πάνω στο κάθε ευρωπαϊκό πλοίο. Αυτό προβλέπεται στην συμφωνία. Αυτά μπορούσα να σας πω ε, εισαγωγικά, προκαταρκτικά. Έχουμε τώρα να κάνουμε με το θέμα της συμφώνου γνώμης του Κοινοβουλίου σχετικά με το πρωτόκολλο αυτό και ελπίζω να μπορέσετε εσείς να δώσετε μια ευνοϊκή γνώμη σχετικά με το πρωτόκολλο αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη αρκετές φορές και επιπλέον όταν εγκρίθηκε πάλι αλλάξε, γιατί κάποιος έλειπε, απουσίαζε. Δεν ρίχνουμε το φταίξιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί φταίμε. Ο κύριος Καπόλας παρακαλώ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας για την ευγένειά σας ε, που συμφωνήσατε να αλλάξετε τη σειρά των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Εγώ σε λίγο θα πρέπει να πάω στο Μεξικό, θα φύγω και δεν περιμένει το αεροπλάνο, βλέπετε, και πρέπει να είμαι στην ώρα μου εκεί. Και ευχαριστώ για την κατανόηση των συναδέλφων. Όπως όλοι γνωρίζουν, πρόκειται για μια μικρή χώρα με τρεις, ε, τρία νησιά που αποτελείται από τρία νησιά βρίσκεται ε, στον Ινδικό ωκεανό πάνω από τον πορθμό της ε, Μοζαμβίκης. Είναι μια μικρή χώρα, μια χώρα που έζησε σε τεράστια πολιτική αστάθεια από τότε που έγινε ανεξάρτητη από τη Γαλλία το 1975. 20 πραξικοπήματα έγιναν από τότε εκεί. Υπάρχει εδώ και η συνιστόσα που είναι σημαντική της ε, βιοτεχνικής αλίας. 30.000 άτομα εξαρτώνται από αυτήν. Είναι μια χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θεσπίσει συμφωνίες αλίας από το 1998. Η τελευταία είναι αυτή που ισχύει τώρα που συνέφθηκε το 2005, τελειώνει του χρόνου 2011, λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ και εξετάζουμε τη νέα συμφωνία, το θέμα της νέας συμφωνίας, που οι γενικότερες σε αδρές γραμμές ε, επεξηγήθηκαν τα θέματα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται για μια συμφωνία που αφορά μικρότερο ποσοστό τόνων, μικρότερο αριθμό τόνων από ότι η προηγούμενη συμφωνία και θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη και την σημαντική ε, αναφορά της Γαλλίας. Ε, τώρα, πέρα από ε, τέτοιου είδους ε, εκθέσεις, για τέτοιου είδους ε, συμφωνίες που θα έλεγα είναι δύσκολος ο συσχετισμός μας αλλά εδώ έχουμε και το θέμα της Επιτροπής όσον αφορά την διαθεσιμότητα, την προθυμία για αυξήσεις, ε, για, για τα έγγραφα. Είχα πολλές δυσκολίες να έχω στη διάθεσή μου τα στοιχεία για να αξιολογήσω ένα τέτοιο θέμα. Φυσικά η συμφωνία αξιολόγησης μόλις την τελευταία στιγμή κατάφερε να καταλήξει σε μια συνθετική παρουσίαση των πραγμάτων. Και δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή διαδικασία με τέτοιες συνθέσεις να καταλήγουμε να αξιολογούμε τα πράγματα όταν έχουμε αξιόλογα θέματα μπροστά μας. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε αλλά δεν θα ήθελα να παραμείνω περισσότερο σε αυτό τώρα. Θέλω στο μέλλον να βελτιωθεί η κατάσταση. Όταν έχουμε τώρα ένα θέμα ε, συμφωνίας αλληλείας ε, θα πρέπει είναι προφανές ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να συμφωνήσει, να μπορεί να συμφωνήσει με τις προτάσεις, διότι πρέπει να αναζητηθούν οι δυνατότητες αλίευσης ώστε να μπορέσουν τα άτομα των ευρωπαϊκών στόλων που δρούν εκεί και αλλιεύουν ένα πολύ σημαντικό αλλιεύμα υπό, υπό ευρωπαϊκής πλευράς στρατηγικής αξίας ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ότι το ποσό αντιστάθμισης είναι σχετικά με, Έχουμε κάπως παραπάνω από 600.000 ευρώ για 70 σκάφη. Να κάνουμε μια τέτοια μικρή σύγκριση, δηλαδή με 1,05% ε, ακριβώς σε ποσοστό ενός ε, ε, τεχνικού που θα παρακολουθεί αυτή την δραστηριότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο, όλο και όλο αυτό έχει ένα πλαίσιο που ε, δίνει κέρδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διαφορετικά πρέπει να πούμε ότι η γραφειοκρατία, το γραφειοκρατικό βάρος είναι υπερβολικό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ανάλογα με το πώς βλέπει κανείς τα πράγματα. Θα ήθελα να θέσω το εξή θέμα. Δεν υπάρχει σε σχέση με την ε, συμμόρφωση, σε σχέση με το 70% της προηγούμενης συμφωνίας για την ανάπτυξη του τομέα της αλληλείας των Κομορών οι ε, εκθέσεις αξιολόγησης αποκαλύπτουν ότι δεν υπήρξε η παραμικρή συμμόρφωση παραμικρή συμμόρφωση σε σχέση με την εφαρμογή κονδυλίων για την ανάπτυξη του τομέα αλληλείας ε, στις ε, Κομόρες. Και εκπλήσωμε περισσότερο όταν παρακολούθησα τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ μεγάλη πίεση όσον αφορά το Μαρόκο μια χώρα που από πλευράς γεωπολιτικής είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρώπη για πολλούς λόγους που δεν θα αναφέρω εδώ και παρακολουθήθηκε από, Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερη θα έλεγα αυστηρότητα ή απαιτήσει όσον αφορά την χρήση των κονδυλίων αυτής της συμφωνίας για την ανάπτυξη ε, στην επικράτεια του Μαρόκου σχετικών δράσεων. Και βλέπουμε ότι κανένα ενδιαφέρον και καμία μέρημνα δεν εκφράστηκε και δεν ελήφθη και το αντίθετο μάλιστα για την ε, από πλευρά της έκθεσης που αφορά τις ε, Κομόρες και για λόγους που δεν ήταν δυνατό να υπάρξει συμμόρφωση με αυτές τις διατάξεις. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει να πιστέψουμε ότι στην επόμενη συμφωνία όπου περίπου το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ε, σκαφών ε, θα ασχολούνται με αυτή την αλληλεία. Και σε σχέση με την έκθεση αξιολόγησης μας λένε ότι εκείνοι που επωφελήθηκαν από τη συμφωνία με τις Κομόρες ήταν οι Σεϊχέλες, η Μαδαγασκάρη, ο Μαυρίκιος, η Νήσος Μαυρίκιος, και ακόμα και η Ταϊλάνδη σε σχέση με τα αλλιεύματα αυτά. Δεν θέλω να ε, προσθέσω άλλα θέματα, Πρόεδρε. Νομίζω σε αυτό το θέμα θα πρέπει να πληροφορηθούμε καλύτερα για τις πραγματικές επιπτώσεις του θέματος και του τι σήμαινε η πειρατεία για την μη, ας το πω έτσι, ε, δυνατότητα, για την ε, κατάσταση των πραγμάτων που δεν έδωσε ευκαιρία να τεθούν τα πράγματα υπό έλεγχο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είμαι πρόθυμος από πλευρά των συναδέφων να ακούσω τις προτάσεις, τις συστάσεις τους και θα τις λάβω υπόψη να είναι δυνατό στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καπόλας. Ε, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Και εγώ από πλευρά μου διεξοδικά, σχετικά διεξοδικά είδα τις αξιολογήσεις για την προηγούμενη συμφωνία και φαίνεται ότι απορρέει από το ότι η παλαιά συμφωνία κόστισε 7,5 εκατομμύρια λέει ευρώ και ότι η αξία των αλλιευμάτων είναι 13,7 εκατομμύρια ευρώ Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ κερδοφόρα η συμφωνία αυτή υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμιά αμφιβόλια με αυτά τα στοιχεία. Αλλά εμείς βρισκόμαστε μπροστά στην μεταρρύθμιση, ενώπιον της μεταρρύθμισης της ε, αλληλευτικής πολιτικής ε, και πρέπει θέματα σαν αυτά να επανεξεταστούν. Γι' αυτό επανεξετάζουμε αυτή τη συμφωνία και επιθυμούμε οι στόχοι μας για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική αλλίας να λαμβάνονται υπόψη. Όπως είπε ο κύριος ε, Καπόλα Σάντος, η αξιολόγηση των προηγούμενων ε, συμφωνιών ε, σε σχέση με την υποστήριξη των τοπικών αλλιέων ήταν κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Δεν πήγε πολύ καλά. Είναι η ίδια ιστορία που ζήσαμε και με τις νήσους Σολομώντα αυτή ότι δεν μπορούσαμε να δούμε πραγματικά να εμφαρμόζονται σωστά οι διατάξεις, ε, οι ε, παράγραφοι για το όφελος των τοπικών αλλιέων. Γιατί δεν έγινε κάποια, ας το πω παρέμβαση για να ληφθούν αυτά τα συμφέροντα υπόψη. Ποιες πρωτοβουλίες λήφθησαν, ώστε νέα μέτρα σε σχέση με τη νέα συμφωνία να, να διασφαλιστούν που θα μπορούσαν με αυτές οι νέες διατάξεις να οδηγήσουν, να κατοχυρώσουν ότι και οι όσοι εργάζονται στα ίδια τα νησιά και δεν είναι αλληλείς και αυτοί να μπορέσουν να υποφεληθούν και οι αλληλείς και οι μη αλληλείς. Γιατί δεν υπήρξαν περισσότερα αλλιεύματα που να έχουν εκφορτωθεί στις κομόρες διότι θέλαμε να υποφεληθούν οι κάτοικοι ε, με την απασχόληση που θα αυξανόταν και γι' αυτό πρέπει οι εκφορτώσεις ε, ε, στις νήσους Κομόρες να συνεισφέρουν τα αλλιεύματα αυτά στην απασχόληση. Γιατί δεν συνέβησαν όλα αυτά λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε. Και η Επιστημονική Οικονομική Επιτροπή Αλίας ανέφερε ότι αυτή η αλία είχε αρνητικές επιπτώσεις για τους, για, για τους γόνους το, του, ε, το, του αλλιεύματος. Υπάρχει υπερβολικά θα έλεγα ε, μεγάλη βλάβη. Είχαμε όμως εμείς δεσμευτεί ότι δεν θα υπήρχε υπεραλίευση από πλευρά τη συμφωνία αλίας που είχαμε συνάψει. Τι γίνεται λοιπόν, δεδομένη αυτή τη αξιολόγηση φαίνεται ότι υπήρξε υπεραλίευση. Και φαίνεται ότι αυτές οι ε, εκτιμήσεις δεν ήταν τόσο καλές όσο εμείς θα το θέλαμε είχαμε εκτιμήσει κάτι το οποίο δεν επετεύθη. Υπάρχει ένας θεός τομέας, θολός τομέας για το τι συμβαίνει. Θα ήθελα να μας τα σχολιάσει όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρος, μάλιστα ευχαριστώ. Κύριε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε εσά θα θέσουμε αυτά τα θέματα, παρότι μπορεί να μην είστε το πιο κατάλληλο να μας απαντήσετε το θέμα. Το θέμα των εκθέσεων αξιολόγησης που ανέφερε ο κύριος Καπόλα Σάντος. Βλέπετε κύριε, εγώ είμαι αναγκασμένη λόγω της θέσεως στην οποία έχουμε καταλήξει τους τελευταίους μήνες, τους τελευταίους μήνες ζητήσαμε να υπάρξει αυτή η αξιολόγηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έστειλε αυτές τις αξιολογήσεις. Έστειλε τις περιλήψεις, συνθετικά τις περιλήψεις των εκθέσεων αξιολόγησης. Και τώρα, σε σχέση με τον αρμόδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του είπα του αρμόδιου δεν μπορούσα να κατανοήσω πώς δεν μας έχει αποσταλεί η πλήρης έκθεση, η πλήρης αξιολόγηση. Και αφού το είχαμε ζητήσει, μας στέλνουν μόνο τις περιλήψεις. Ε, σε, μέσα σε μια νύχτα αυτά από τη μια μέρα στην άλλα, άλλη έγιναν λέει απόρριτα, εμπιστευτικά θέματα και δεν μπορούσαν λέει να μας αποκαλυφθούν προηγούμενα δεν υπήρχαν προβλήματα. Τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και με τις καλές σχέσεις που υποτίθεται ότι αναπτύσσονται μεταξύ των, οργάνων της Ένωσης, τώρα δεν μας αποστέλουν αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης. Μπορεί κάποιος να μας επεξηγήσει γιατί αυτό έχει γίνει εμπιστευτικού χαρακτήρα θέμα ή απόρριτο τώρα τελευταία. Και εγώ είμαι πεισμένη Είμαι βέβαιος ότι, βεβαία ότι για αυτόν τον τομέα ως ε, Ευρωβουλευτήνα, ως Πρόεδρος δεν μπορώ να ε, βασιστώ σε φήμες. Τα τελευταία που μας είχαν αποσταλεί ήταν σε σχέση με την έκθεση για την οποία ήμουν αρμόδια. Αλλά εδώ έχουμε τον Ιούνιο που ήταν τότε. Τον τελευταίο όμως καιρό και για τις νήσους Σεϊχέλες, Κομόρες δεν μας δίνουν τα πλήρη στοιχεία αλλά μόνο περιλήψεις. Συνθετικέ περιλήψει. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσεί με του δικού σα, αλλά εγώ θέλω να εκφράσω δημόσια το παράπονο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση χωρί να έχουμε τι εκθέσει αξιολόγηση, Γελιοποιούνται τα πράγματα κιόλα ξαφνικά. Από τη μια μέρα στην άλλη μα λένε ότι είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα αυτά τα στοιχεία. Ποια είναι η λογική πίσω από όλα αυτά. Δεν το κατανοώ. Τώρα τούτων λεχθέντων αυτό εκρεμεί ακόμα εκρεμεί και πρέπει να επιληθεί με κάποιο τρόπο. Διότι πραγματικά είναι αλήθεια, δεν ξέρω γιατί δεν είναι δυνατόν να δουλέψουμε όπως πρέπει και όπως είναι ε, ανάγκη να δουλέψουμε σωστά με τα στοιχεία που είναι αναγκαία να έχουμε στα χέρια μας. Και για κάθε ευρωβουλευτή επιπλέον, όχι μόνο για μένα, όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον αυτό είναι δεδομένο και πρέπει να μπορούν να τα διαβάσουν, αλλά δεν είναι στη διάθεσή τους. Και τώρα είναι το θέμα του συστήματος και τη μεθόδου εργασίας πρέπει να μας απασχολήσει. Αλλά περνάμε στο θέμα τώρα των κομορών, κύριε. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Αληθεύει αληθεύει ότι κατά, ε, το πέρασμα των ε, παραγαδιάρικων από το 2007-2008 υπήρχε 98% ε, χρήση, εκμετάλλευση, εξάντληση των δυνατοτήτων αλίας. 98% ίσον 100% δηλαδή. Αληθεύει ότι το 2009 και 2010 μειώθηκε η απόδοση λόγω πειρατείας και αυτό είναι, αναφέρεται και από την περίληψη της έκθεσης αξιολόγησης. Πράγμα που είναι λογικό γιατί έχουμε την περιοχή εκεί κοντά στη Μαδαγασκάρη και έχουμε και το θέμα της ε, πειρατείας. Λοιπόν, για την αύξηση των ε, παραγαδιάρικων που μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι ίσως αυτό θα ήταν ε, δικαιολογημένο, είχαμε 27 πριν με, τους, με, τα σειρώμενα δίκτυα και τώρα έχουμε 25. Και αυτό δεν συμπίπτει ακριβώς με την πειρατεία. Πώς μπορείτε να μας εξηγήσετε ότι είχαμε αύξηση σε 25 όταν είχαμε την ε, ε, χρήση για τα ε, όσα σέρνουν δίκτυα σε 24. Υπάρχει κάποιος λόγος που μπορεί να εξηγήσει αυτή την κατάσταση. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι της τομεακής υποστήριξης, της κλαδικής ή τομεακής υποστήριξης. Η Επιτροπή το 2008 είχε πει ότι πράγμα το οποίο είναι επαναληπτικό σε όλες τις συμφωνίες αλίας ότι δεν υπήρξαν μεγάλες πρόοδοι όσον αφορά την τομεακή υποστήριξη. Γι' αυτό με εκπλήσει ότι τώρα πάλι υπάρχει μια τόσο μεγάλη ποσότητα, 300.000 ευρώ, για την τομεακή υποστήριξη. Όταν έγιναν τόσα λίγα λέγεται στο παρελθόν. Πολύ δύσκολα μπορώ να θεωρήσω ότι δικαιολογείται να περνάμε σε τέτοια ποσά ετήσια 315.000 ευρώ για την αντιστάθμιση επειδή υπήρξε λέει μείωση των δυνατοτήτων αλληλείας αλλά 300.000 για τον τομέα αυτόν την τομεακή υποστήριξη όταν δεν έχει γίνει τίποτα δύσκολα μπορεί να το καταλάβει κανείς. Όταν επιπλέον το παράπονο το οποίο είχε διατυπωθεί είναι ότι δεν έχουν ε, ε, δεν έχουν υποστήριξη για να προχωρήσει η τομεακή ανάπτυξη. Είναι ένα θέμα λοιπόν αυτό που θα έπρεπε να αλλάξουν οι σχέσεις και ο συσχετισμός με, την, ε, με τα νησιά Κομόρες γιατί δεν έχουν ε, το υλικό και το δυναμικό για να μπορέσουν να αναπτύξουν τομεακά αυτόν τον τομέα. Και υπάρχει ένα θέμα τώρα εδώ για την ε, ναυτολόγηση ναυτικών σε σχέση με την Μικτή Επιτροπή. Αυτά τα σκάφη, οι Κομόρες δεν έχουν λιμάνια, επαρκή λιμάνια, εφοδιασμένα επαρκώς λιμάνια για να πάνε εκεί τα πλοία μας και να εκφορτώνουν εκεί. Το μόνο λιμάνι που λειτουργεί εκεί πέρα από τη Μαδαγασκάρη είναι η, η ΜΑΕ των Σεϊχελών, η, η Βικτόρια, η πρωτεύουσα των Σε, ε, Σεϊχελών νήσων. Δεν έχουν τις ελάχιστες υποδομές οι κομόρες, ώστε τέτοιου είδους ε, αλλιευτικά να μπορούν να, να εκφορτώνουν εκεί. Ίσως γι' αυτό έχουμε και πρόβλημα για την αυτολόγηση ε, ναυτικών. Αν δεν μπορεί να φτάσει εκεί κάποιο ε, σκάφος ε, να ξεφορτώσει, δεν μπορούν να ναυτολογηθούν εκεί κιόλας ναυτικοί. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να ναυτολογηθούν χωρίς να μπορούν να προσεγγίσουν λιμάνια στις Κομόρες τα, σκάφη. Θα ήθελα να μου τα εξηγήσετε όλα αυτά για να τα κατανοήσω. Η κυρία Μπιλμπάο μετά από αυτό, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω με τα θετικά. Η ανανέωση οποιασδήποτε συμφωνίας, όπως έχουμε και αυτή μπροστά μας, είναι μια συμφωνία που είναι υπέρ των ε, σκαφών της Ευρώπης που αλλιεύουν εκεί και είναι κάτι θετικό για μας. Με το πέρασμα των ετών, καθώς περνάει ο χρόνος, τα αρνητικά στοιχεία εκείνα πέρα από αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, έλλειψη πληροφόρησης ε, σε σχέση με τα μέλη της Επιτροπής Αλληλείας, με αυτές τις εκθέσεις που δεν μας δίνονται και δεν έχουμε στα χέρια μας ε, και απουσία έλλειψη στοιχείων αριθμητικών και άλλων, θα ήθελα να μπορούσαμε να τα αναλύσουμε αυτά και σε σχέση με τον έλεγχο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πάντα δημιουργεί ερωτηματικά όταν αλλιεύει υπό ευρωπαϊκές συμφωνίες ο Ευρωπαϊκός Τόλο εκεί, θα ήθελα να ξέρω, εσείς συντάξατε κάποια έκθεση για την ενσωμάτωση σε αυτή τη συμφωνία του θέματος του ελέγχου, των ελέγχων που γίνονται για τις, ε, την αλλιευτική δράση των ε, ευρωπαϊκών σκαφών και υπό τις προηγούμενες συμφωνίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ζητήσω και σε σχέση και με, το, με τα σκάφη ε, που αλλιεύουν τόνο. Αναφέρθηκε ότι αλλιεύουν παράνομα, αλλιεύουν εκεί που δεν έπρεπε να βρίσκονται. Με ενδιαφέρει, έχετε αναλύσει όλα αυτά τα φαινόμενα εσείς ή όχι ώστε να μπορέσουμε να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία με καθαρή συνείδηση. Αν δεν το κάνετε, έχετε προβλέψει ότι θα το κάνετε και μετά σε σχέση με τη συμφωνία, για να μην επαναλάβω πράγματα που προαναφέρθηκαν, εσείς κάνετε λόγο για τις νέε δυνατότητε αλληλεία. Όταν κάνετε λόγο για νέε δυνατότητε αλληλεία, κάνετε λόγο για την προαγωγή της ε, πειραματικής αλίας και αν αυτή η πειραματική αλληλεία θα μπορούσε να ενταχθεί και να διευρυνθεί υπό αυτή τη συμφωνία. Σας ερωτώ, έχετε υπόψη κάτι εξειδικευμένο και συγκεκριμένο για αυτή την εξαντλητική, ας το πω έτσι, ε, τοποθέτηση ή ε, δράση για τα ε, θηνοειδή, για παράδειγμα, που είναι και άλλο θέμα και στο ε, δάφιο 2, στο άρθρο 2, γίνεται λόγος για τις πιθανές, τα πιθανά λιεύματα και το τι θα έπρεπε να πληρώσουμε εμείς ως αντιστάθμισμα γι' αυτό. Κάντε λόγο και για την δυνατότητα αύξησης των αλλιευμάτων, το διπλάσιο κιόλα αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν αντιβαίνει, δεν αντιφάσκει με τα στοιχεία της ΕΚΑΤ που κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ε, είχαν ε, συγκροτηθεί, είχαν θεσπιστεί ουσιαστικά ίσως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσα θα μπορούσαμε να αλλιεύουμε αλλιεύματα σε, αυτές, σε αυτές τις ζώνες. Θα ήθελα να μου απαντήσετε αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα ερωτήματα που ετέθησαν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο δυνατόν καλύτερα και ίσως να απευθυνθώ και στη συνάδελφο που είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο θέμα για να συμπληρώσει απαντήσουμε, αν μου επιτρέπετε. κατόπιν της παρουσίας που θα κάνω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας κάποια πράγματα πάνω στη γενική εισαγωγή σας ό,τι αφορά την ε, ε, μεταβίβαση των εκθέσεων αξιολόγησης. Παρακαλώ πολύ δεχτείτε ότι δεν είμαι υπεύθυνο και υπόλογος του θέματος αυτού. Απλώς πληροφοριακά θα ήθελα να σα εξηγήσω αυτό που ίσω αν θέλετε να έχει νόημα και ένα λογικό στο έγγραφο αυτό και που ίσω επεξηγεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτέ οι αξιολογήσει άπτονται κάποιων κρίσεων σε ό,τι αφορά την εσωτερική διοίκηση των τρίτων χωρών αφορούν σε χρηματοοικονομικά θέματα, σε αναλύσεις προπολογισμών, δημοσιονομικές αναλύσεις. Είναι αρκετά ειλικρινή σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική κατάσταση των χωρών αυτών όταν βεβαίως καταφέρουμε να βρούμε πληροφορίες ε, με την, και ενδεχομένως με κατόπιν συμφωνίας με τρίτες χώρες. Είναι στοιχεία λοιπόν τα οποία αν μη τι άλλο οι τρίτες χώρες θεωρούν αυτές κατά αυτές ότι είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στοιχεία. Αυτή ήταν η μόνη πληροφορία που μπορούσα να σας δώσω σχετικά. Τα υπόλοιπα βέβαια τίθεται σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο που μου εκφεύγει πλήρως, ε, όπως πολύ σωστά επισημάνατε και εσείς. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία αυτή με τις Κομόρες, ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προηγούμενη συμφωνία δεν κάλυπτε αυτή τη διάκριση που υπάρχει σήμερα σε όλες σχεδόν τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης που έχουμε συνάψει και που κάνουν ακριβώς διάκριση μεταξύ του ποσού το οποίο θα διατεθεί για την πληρωμή για να υπάρξει πρόσβαση στην πηγή αφενός και του τμήματος της συνεισφοράς που προορίζεται στην ε, υποστήριξη της ε, ΚΑΠ. Η νέα αυτή συμφωνία λοιπόν εισάγει αυτή τη διάκριση κατά τρόπο απόλυτα σαφή. Είναι ελθές ότι οι κομόρες αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να εφαρμόσουν αυτά που είχαν προβλεφθεί στην, ε, στα σχετικά της ε, ενίσχυσης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Είναι μια εξαιρετικά φτωχή χώρα, εξαιρετικά φτωχή, της οποίας ε, η διοίκηση ορισμένε φορές είναι πραγματικά στοιχειώδης και που χρήζει πολύ μεγάλες ε, βοήθειες. Θα έλεγα ότι η διαφορά μεταξύ των Κομορών και, ε, του Μαρόκου, γιατί αναφέρθηκε προηγουμένω, είναι ότι το Μαρόκο έχει μια εξαιρετικά ικανή και ε, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, που έχει και ίδια αλλιευτική πολιτική και επομένως από την οποία δημόσια διοίκηση μπορούμε να ζητήσουμε λογαριασμούς και εκθέσεις με πολύ πιο ενεργητικό τρόπο παρά από μια χώρα όπως οι Κομόρες που είναι μια από τις πλέον φτωχές της περιφέρειας με την οποία έχουμε μια συμφωνία τέτοιου τύπου. Αυτό δεν με οδηγεί να σας πω ότι ακριβώς αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ε, θελήσαμε και επιθυμήσαμε να αυξήσουμε το κομμάτι της συμφωνίας το οποίο πρόκειται να υποστηρίξει την πολιτική αλίας χάρη νομίζω αν μη τι άλλο εν μέρη της συμφωνίας αυτής οι Κομόρες έχουν ε, χάρη της συμφωνίας αυτής μια πολύ ικανή ε, διοίκηση ό,τι αφορά την Αλία που επέτρεψε στη χώρα αυτή να ε, συνδράμει πολύ ενεργητικά στο περιφερειακό πρόγραμμα Αλίας στην περιοχή του Ινδικού και να εγκατασταθεί στις Κομόρες ένα κέντρο επιτήρησης, παρακολούθησης, το οποίο συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια εποπτείας επιθεώρησης της αλίας. Μιλάω αμυγός εποπτεία για την αλία, για κάτι άλλο. Οι κομόρες λοιπόν συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα επιτήρησης και επιθεώρησης της αλίας στον Ινδικό ωκεανό και μπορούμε να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουμε για την υποστήριξη της χώρας αυτής. Αυτά σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, γιατί ετέθη το ερώτημα και στα θέματα ελέγχου. Νομίζω ότι ο ειδικό Οικιανό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε, υποστηρίζοντα τι προσπάθειε αυτέ τη ίδια τη χώρα, που προσπαθούν σε συγκερασμό των δυνάμεών του για να μπορέσουν να επιτηρήσουν τον τεράστιο χώρο, την τεράστια περιοχή στην οποία, διαπλέουν την οποία διαπλέουν ε, πει στόλοι, μεταξύ των οποίων και δική μα. Αυτά σε ό,τι αφορά τις εκφορτώσεις, σε ό,τι αφορά τις εκφορτώσεις τώρα. Προφανώς δεν υπάρχει διαθέσιμη υποδομή σήμερα στις κομόρες για αυτές τις εκφορτώσεις. Και ένα κομμάτι της αρρωγής που την οποία διαθέτουν θα μπορούσε ακριβώς να βοηθήσει τη χώρα αυτή να αποκτήσει αυτή την ελάχιστη υποδομή που θα της επέτρεπε να διαδραματίσει πολύ ενεργό ρόλο σε αυτό που συμβαίνει στην ε, αρχή της ε, Τη ε, αλυσίδα αυτής, δηλαδή την αρχική επεξεργασία των αλλιευμάτων. Αυτή τη στιγμή τα αλλιεύματα κατά κύριο λόγο ε, προωθούνται στις Σεϊχέλε, όπου γίνεται μια πρώτη επεξεργασία. Δεν κατάλαβα την αναφορά στην ΙΚΑΤ που έγινε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους γόνους. Η Επιτροπή αυτή δεν έχει τίποτα να κάνει, γιατί η ΚΑΤ καλύπτει το Ατλαντικό και Μεσόγειο. Γιατί αναφέρθηκε. Εκτός μικροφώνου η παρέμβαση. Σε ό,τι αφορά τους γόνους, δεν αναφέρθηκα στην ΕΚΑΤ, αναφέρθηκα στην ε, STSF. Συγγνώμη, λάθος μου τότε. Συγγνώμη, συνεχίζω στα γαλλικά. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στα θέματα των γόνων, στην ΙΚΑΤ για τον τόνο, αλλά εδώ μιλάμε για λιεύματα ανοιχτά τη Αφρική και πιο συγκεκριμένα στον κόλπο τη Γουινέα. Και το συζητήσαμε αυτή τη βδομάδα. Αλλά όντως η ε, γόνοι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η αρμόδια επιτροπή για τον Ειδικό ωκεανό και που ε, εκδίδει τους σχετικού κανόνε είναι η Επιτροπή του Ειδικού Ωκεανού για την Αλία του Τόνου, η IOTC στα αγγλικά και η οποία καθορίζει την ε, κατάσταση των αλλιευμάτων που αναφέρει ότι είναι ανησυχητικά για κάποια είδη και δει για παράδειγμα για τον κίτρινόπτερο τόνο είναι πολύ καλύτερα για τον ε, ερθρό που αλλιεύεται στα ανοιχτά του Ινδικού και στον Ειρηνικό ωκεανό. Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα των ε, παραδιών, παραγαδιάρικων και των μεγάλων, όντως έχουν πληγεί από την πειρατεία, πράγμα που έχει οδηγήσει σε μια μετατόπιση αυτής της αλληλευτικής δραστηριότητας προς τον Ατλαντικό, πράγμα το οποίο μας ε, ανησυχεί οι, οι ευρωπαϊκοί στόλοι έχουν καταφέρει να ενταχθούν με αρμονικό τρόπο ε, και να προσαρμοστούν στις υφιστάμενες δυνατότητες αλίευσης, αλλά βλέπουμε να φτάνουν πάρα πολλά πλοία από την Ταϊβάν και από την Κορέα στον Ατλαντικό, που ακριβώς εκφεύγουν των ε, ζωνών αλίας του Ινδικού ωκεανού λόγω της ε, προεξάχουσας πειρατείας. Ε, το θέμα της πειρατείας δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά τα οποία δεν είναι ήδη γνωστά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι αλλοίς να τύχουν κάποιες προστασίες που αυτή τη στιγμή εστιάζει κατά κύριο λόγο στα μεγάλα εμπορικά πλοία. Είναι σημαντικό όμως να προστατευτούν με τον ίδιο μηχανισμό και οι αλλοίς. Είναι αναγκαιότητα. Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις τελευταίες προφορίες που έχουμε λάβει, τα ευρωπαϊκά πλοία είναι πολύ συχνά θύματα επιθέσεων ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Τα περισσότερα από τα πλοία, αυτή, τα, από τα πλοία αυτά σήμερα ε, προστατεύονται σε ό,τι το γαλλικό στόλο από στρατιωτικές δυνάμεις. Στην περίπτωση των ισπανικών πλοίων από, τις, ε, από ιδιωτικές μυστικές υπηρεσίες, ε, από ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, εν λόγω περιοχή ενδιαφέροντος αλλία, τις Κομόρες δηλαδή, είναι μια περιοχή που εστιάζει στον τόνο, που είναι ένα είδος βέβαια εξαιρετικά μεταναστευτικό. Είναι σημαντικό οι αλλιευτικές ζώνες ε, να είναι ως το δυνατόν πιο καλά περιχαρακωμένες για να μπορούν να, ε, να υπάρχει έλεγχος σχετικής αλίας. Τα αποθέματα σύμφωνα με την εποχή και τις περιβαλλοντικές συνθήκες θα μετατίθενται και να το πείτε από τη μία ζώνη στην άλλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η ελία θα είναι εξίσου παραγωγική από τη μία χρονιά στην άλλη. Αυτές οι αλληλευτικές συμφωνίες λοιπόν, και πρέπει να υπογραμμιστεί αυτό, είναι συμφωνίες οι οποίες επιτρέπουν να καθορίσουμε ένα ελάχιστο ποσό πρόσβασης στην αλίευση. Μπορεί όμως να συμβεί αυτή η πρόσβαση στην αλίευση να μην χρησιμοποιείται ορισμένε φορές και να μην εξαντλείται από τους ευρωπαϊκούς τόλους, από τα ευρωπαϊκά πλοία. Ετέθη ένα ερώτημα πάνω στα παραδιάρικα, καθώς και τις νέες δυνατότητες αλίες στην περιοχή. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο, η οποία μπορεί να απαντήσει με μεγαλύτερη, περισσότερη ακρίβεια. Ευχαριστώ. Σχετικά με τις αλλιευτικές δυνατότητες, οι οποίες περιγράφηκαν, υπάρχει δυνατότητα για τους εφοπλιστές να έχουν ένα δίκτυο δραστηριοτήτων στην ε, διάθεσή τους για να μπορούν να κάνουν προβλέψεις. Αυτό όμως δεν είναι τόσο εύκολο για τα παραγαδιάρικα όπως ε, για τα πλοία με γρηγρή, ε, τους γρήπους, διότι τα παραγαδιάρικα πλοία είναι δυσκολότερο να να επιτρέψουν προβλέψεις. Γι' αυτό οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και των εφοπλιστών μας επιβιώνουν κάθε φορά την δυνατότητα να διατηρήσουν τις δυνατότητες με τα παραγαδιάρικα, γι' αυτό εισήχθηκαν ε, αντικατοπτρίζοντας τα αιτήματά τους όπως και τις ε, δυνατότητες ε, αλίευσης με την κατηγορία των πλοίων με γρηγρή όπως και με την Γαλλία που προκύπτει από ένα νέο σχέδιο, ένα νέο ε, πρόγραμμα με τα όρια που έχουν επιβλωθεί από την ε, Επιτροπή για τα Αθηνοειδή του Ινδικού Ωκεανού που έχει αρμοδιότητα στον τομέα αυτών. Τούτων λεχθέντων θα ήθελα επίσης ε, να αναφερθώ και στους ναυτικούς από τις Κομόρες που επισημάνθηκε Βεβαίως οι διατάξεις, οι τεχνικές ε, και οι πρακτικές ε, θα εφαρμοστούν. Έχουμε αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα για να επιτρέψουμε να υπάρξει ένας ναυτικός από τις Κομόρες σε κάθε πλοίο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα αυτή. Η χώρα αυτή έχει καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες οικονομικές για να επιτρέψει την εκπαίδευση και κατάρτιση 15 πλοιάρχων αλλιευτικών πλοίων ε, που εκπαιδεύτηκαν στην σχολή Μαϊάγκα κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Έχουν λοιπόν επενδύσει στην κατάρτιση αυτών των ατόμων και θα πρέπει και εμείς ε, να τηρήσουμε την διάταξη αυτή στον τομέα αυτών και να διατηρήσουμε αυτόν τον τοπικό ιστό που υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε τις πρακτικές ρυθμίσεις και διευθετήσεις στην επόμενη μικτή επιτροπή, οι οποίοι θα, τις οποίες θα προηγηθούν τεχνικές συνεδριάσεις, ούτως ώστε να προβλέψουμε μια, ένα πλαίσιο για να μπορούμε να, να προσδιορίσουμε όλες τις δραστηριότητες του τομέα που αναφέρθηκαν επίσης για να επιτρέψουμε μια ανάπτυξη, η οποία υπάρχει ήδη χάρη στους πόρους που διατέθηκαν ήδη στα πλαίσια του Περιφερειακού Προγράμματος Παρακολούθησης της Αλίας. Γι' αυτό οι κομόρες μπόρεσαν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και τις δυνατότητές τους που τους επιτρέπουν να έχουμε περισσότερα μέσα για να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο στον τομέα αυτών. Κυρία Πρόεδρε, απλώς να προσθέσω κάτι για να κλείσω και να σας δώσω μια ιδέα του μεγέθους της σημασίας της εργασίας που απομένει ακόμα να γίνει με αυτήν την αναπτυσσόμενη χώρα. Οι κομόρες δεν έχουν ποτέ υποβάλει στοιχεία αξιόπιστα ε, στην CTOE. Ε, θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουν ε, να συλλέξουν στοιχεία στατιστικά. Είναι όμως μια χώρα η οποία έχει όμως ένα νόμο πλαίσιο για την αλληλεία είναι μεγάλη ε, πρόοδο το ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο το ε, επιχειρησιακό, το πολιτικό. Πιστεύω λοιπόν ότι η αύξηση η οποία δόθηκε στη χώρα αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας αυτής που είναι τεράστιες και θα πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή για να μπορέσει να αναλάβει ε, την ευθύνη της ε, στην διακυβέρνηση της Αλίας σε αυτήν την περιοχή του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι απήντησα περίπου στο σύνολο των ερωτήσεων που μου τέθηκαν. Η κυρία Ανδρές Μπαρέα θέλει να διατυπώσει μια ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξειδικεύσει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκθέσεις αξιολόγησης που ανέφερε ότι καταδείχθηκε ότι είναι περιορισμένες τώρα, είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα για την δημοσιονομική ανάλυση και οικονομική ανάλυση για τα θέματα αυτά. Η απάντηση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν, είπε ότι αυτό οφείλεται στην μη ικανότητα, διοικητική ικανότητα να ανταποκριθούν στη διάθεση αυτών των στοιχείων τα νησιά Κομόρες. Θέλω να πω ότι δεν είναι ανικανότητα διοικητική, είναι προφανές ότι η μη ικανότητα από διοικητικής πλευράς θέτει προβλήματα, ότι η έλλειψη ανάπτυξης διοικητικά είναι προφανής, όμως ευαίσθητα στοιχεία οποιασδήποτε, οποιασδήποτε χώρας ή οποιοδήποτε φορέα ή οργάνωσης για το ότι μπορεί εδώ να μπορούν να αλλοιωθούν, να αλλάξουν κάποια στοιχεία είναι κάτι διαφορετικό. Δεν εξαρτάται από την διοικητική ικανότητα, το να φτάσουμε σε κάποιο σημείο συμφωνίας. Γιατί δεν αποστέλλονται οι πλήρεις εκθέσεις. Το να είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα σημαίνει περιορισμένη ε, ε, ε το πω έτσι, η διάθεση. Το να υπάρχει όμως διοικητική ανικανότητα είναι άλλο θέμα. Γιατί το ένα είναι εμπιστευτικό λοιπόν και γιατί εσείς επικαλείστε θέματα μη ικανότητα διοικητικής των κομωρών ίσων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και μας αφορά εμάς. Ε, κύριε Λόβε, παρακαλώ. Sorry, I Συγγνώμη. Ήθελα μόνο να ρωτήσω και πάλι. Ε, να επανέλθω. Εκτιμώ αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ανάγκη των κομωρών να δημιουργήσουν υποδομές και να αναπτύξουν τη δική τους αλληλευτική πολιτική. Δεν καταλαβαίνω όμως πώς αυτή η νέα συμφωνία θα εξασφαλίσει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποιες ε, νέες συνιστώσεις στη συμφωνία αυτή, που θα προβλέπουν μια παρακολούθηση και την επιτόπου ε, αρρωγή στις κομόρες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο εκπρόσωπος Επιτροπής. Ευχαριστώ που μου υπενθυμίσατε, και πάλι ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνο τη Γενική Αλλιευτική Πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση των εγγράφων και των εκθέσεων. Προσπάθησα μόνο να πληροφορήσω την Επιτροπή σα στο τι θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ευαίσθητε πληροφορίε τη εκθέση αξιολόγηση. Όμως ε, είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσουν σε ό,τι αφορά την επεξεργασία και τη μετώπιση αυτών των, των εβέστων, λόγω ευαίσθητων πληροφοριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη νέα προσέγγιση με τη νέα προτινόμενη συμφωνία ε, για την ε, υποστήριξη και την εφαρμογή μιας βιώσιμης αλληλευτικής πολιτικής, Καταρχά, θα πρέπει να αναγνωριστεί και να εντοπιστεί ένα συγκεκριμένο ποσό, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στην προηγούμενη συμφωνία. Στο παρελθόν, αν θέλετε, ήταν μια παλιά πρακτική που χρησιμοποιείται. Σήμερα υπάρχει ένα σαφέστατο ποσό για τι δραστηριότητε αυτέ. Αυτό είναι το πρώτο καινούριο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο, σύμφωνα με ό,τι γίνεται και με τι άλλε συμφωνίε, θα υπάρχει μια ε, μήτρα, αν θέλετε, που απορρέει από που είναι το προϊόν συζητήσεων μεταξύ του ε, υποψήφιου ε, ευεργετούμενου κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που επιτρέπει να καθοριστούν σαφώς οι, στόχοι ανάπτυξης. Αυτή η μήτρα, θέλετε, θα αποτελεί αφενός με ένα πρόγραμμα εργασίας για τις κομόρες και αφετέρου έναν τρόπο εξασφάλισης της παρακολούθησης των εκταμιεύσεων και της πρόοδου των διαφόρων ε, έργων. Υπάρχει λοιπόν ένας κοινός ορισμός των μεγάλων στόχων που τίθενται σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ε, χώρας και τουλάχιστον στα πλαίσια της κοινή Επιτροπής, αλλά και κατά τη διάρκεια των τεχνικών επιτροπών, θα δοθεί δυνατότητα να επανεξεταστούν μαζί με τις ε, υπεύθυνου των κομορών την πρόοδο αυτή της ε, πτυχής συνεργασίας μας. Νομίζω λοιπόν ότι υπό αυτή την έννοια θα έχουμε μια πολύ καλή παρακολούθηση και κάτι καλύτερα δομημένο σε σχέση με αυτό που είχαμε μέχρι τώρα με την χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Gracias, señor ponente. Ε, σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Καπόλα Σάντος. Ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις και προτάσεις. Δύο παρατηρήσεις. Το άρθρο 7 του πρωτοκόλου, του προηγούμενου πρωτοκόλου, αντιφάσκει απόλυτα με αυτά τα οποία μόλις ακούσαμε. Λέει ακριβώς ότι 60% των προηγουμένων κονδυλίων έπρεπε να είχαν δοθεί στην ανάπτυξη του τομέα της αλληλείας. Και το λέει αυτό με απόλυτα σαφή τρόπο. Η άλλη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξή. Είναι κρίμα κρίμα ότι εμείς ε, παρεμβαίνουμε μόνο στην φάση όταν όλα έχουν πλέον ε, εκτελεστεί και έχουν γίνει. Εμείς να πούμε ναι ή όχι, να εγκρίνουμε ή να καταψηφίσουμε. Και ποτέ φυσικά να πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Στόλο Αλίας δεν θα πούμε όχι. Αλλά πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε κάτι. Προτού είναι τελεσίδικα τα πράγματα πια. Προτού είναι η τελευταία φάση και έχουν όλα γίνει και είναι συντελεσμένα. Για να μπορέσουμε κάπως να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των κομορών που είναι η κύρια, το κύριο εμπόδιο για να μπορέσει να αποκομίσει ωφέλη από την αλία στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είναι ανώφελο, δεν μπορεί να γίνει κάτι για, απλά θέτω αυτή την ε, πτυχή στην έκθεσή μου για ιστερότερες συμφωνίες και θέλω να ολοκληρώσω ζητώντας συγγνώμη από τους συναδέφους για τη δυσκολία που προκάλεσα έχοντας αλλάξει την ημερήσια διάταξη λόγω των ανηλυμένων υποχρεώσεών μου. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Eh, Μόνο ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω λέει η Πρόεδρος. Προσπαθούμε με τις συνθήκη της Λισαβόνας να αλλάξουμε ακριβώς όλη αυτή τη διεργασία, τη διαδικασία σε σχέση με συμφωνίες αλληλείας και να εμπλεκόμαστε έγκαιρα ως κοινοβούλιο σε αυτά τα θέματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναφέρει. Είναι αδύνατο λοιπόν ε, ιστερότερα να, έχει, να μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Και Επίση, θα πρέπει να αποσαφινιστεί η διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη διάθεση των ε, ε, εκθέσεων αξιολόγηση. Είχαμε χρόνια ολόκληρα τέτοιου είδου εκθέσεις στη διάθεσή μα τώρα εξαφανίζονται, δεν μας διατίθενται πλέον. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Θα πρέπει να δούμε πώς θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα, διότι εκρεμεί και πρέπει να επιληθεί. Δεύτερο, δεύτερο, μια στιγμή. Λοιπόν, κατά δεύτερο λόγο, είναι αλήθεια αυτό το οποίο αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Είναι δύο τμήματα τώρα ξεχωριστά. Είχαμε ένα ξεχωριστό ποσοστό πιο πριν, το οποίο στόχευε για την τομεακή ανάπτυξη. Τώρα έχουμε δύο διαφορετικά σκέλη και είναι διαφορετικό το ένα με το άλλο σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Νομίζω σωστά καταβάλλονται οι προσπάθειε, αλλά πρέπει να γίνει κάτι και με το λιμάνι για ένα λιμάνι στι Κομόρες για τι υποδομέ. κάτι πρέπει να γίνει στις μικτές ε, επιτροπές αντιπροσωπείες ε, ένα πρόγραμμα που υποβάλλει μια τρίτη χώρα μετά ε, γίνεται αντικείμενο διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορούν να τεθούν κάποιοι προσανατολισμοί αλλά δεν μπορούν να επιβληθούν σε μια τρίτη χώρα το να γίνει λοιπόν ένα λιμάνι στι Κομόρες που όλοι γνωρίζουμε να, ότι είναι χρήσιμο ως πλατφόρμα κτλ. Λοιπόν, ολοκληρώνω. <clears throat> Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, μπορεί να εξεταστεί αν είναι προτεραιότητα, αν πρέπει να γίνει ένα λιμάνι στις Κομόρες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπεται και σε σχέση και με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, παρουσίαση της έκθεσης. Παρουσίαση της έκθεσης 25-26 Ιανουαρίου ψήφιση στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή στη συνάντηση του Μαρτίου. Στην Ολομέλεια θα περάσουμε στην Ολομέλεια του Απριλίου. Αυτά έχουν προβλεφθεί από πλευρά χρονοδιαγράμματος. Λοιπόν, προχωράμε αμέσως, ολοκληρώνεται αυτό το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστούμε τον κύριο Καπόλα Σάντος για το έργο που έκανε. Και τώρα περνάμε στο 7 της ημερήσιας διάταξης τροποποίηση του κανονισμού της Ευρωπαϊκή, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1288 2009 σε σχέση με την θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων από το 2011 έως τις 30 Ιουνίου 2011. Η ε, κυρία Γκρεντιέ Αρμόδια ήταν υπεύθυνη, η συγγήτρια, η κυρία Γκρεντιέ, θα μας ε, κάνει την, την παρουσίαση της έκθεσής της. Έχετε τον λόγο κυρία Γκρέντια, παρακαλώ. Madame la Présidente. Κυρία Πρόεδρε, το αντικείμενο αυτής της έκθεσης είναι το αίτημα της Κομισιόν ε, να παρατείνουμε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013 την ισχύ ε, του κανονισμού που αναφέρεται στις μεταβατικές ε, τεχνικές, τα μεταβαστικά τεχνικά μέτρα τα οποία ε, έπρεπε να λήξουν στις 30 Ιουνίου 2011. Έχει παραταθεί, πρόκειται για έναν κανονισμό του 2008 λόγω της ε, αδυναμίας να συμφωνήσουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σήμερα το πλαίσιο είναι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες εκθέσεις αλλαγής διαδικασίας από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Έχουμε ενισχυμένο ρόλο εμείς στο Κοινοβούλιο και θέλουμε να συμμετάσχουμε στην συζήτηση, αλλά κυρίως μέσα στην προοπτική της μεταρρύθμισης της κοινή αλλιευτικής πολιτικής ε, και την πρόταση που περιμένουμε από την Επιτροπή στα μέσα του 2011 και που θα πρέπει να εντάξει αυτά τα τεχνικά μέτρα. Ζήτω λοιπόν να απαντήσουμε στο αίτημα της Επιτροπής χωρίς σημαντική αλλαγή με μόνο μια διευκρίνηση ε, νομική, απλώς να διευκρινίσουμε ότι τα ενδιαφερόμενα κρατημέλη θα υποβάλλουν ε, στην Κομισιόν. Αυτό δεν αναφερόταν ε, στο αρχικό κείμενο, αλλά κυρίως πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή ότι η περίοδος παράτασης αυτού του κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις ε, πάνω στα πλοία και στα οικοσυστήματα, όπως είχε αναλάβει η Επιτροπή και υποστηρίζω την πρόταση που έγινε από τον συναδελφό Γκάλαγκερ στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε σχετικά με την έκθεση αυτή για την πρόσκληση που απευθύνατε εσείς κυρία Πρόεδρε και τα μέλη της Επιτροπής για τα συμβούλια τα περιφερειακά να έρθουν να μας παρουσιάσουν επιπτώσεις των μέτρων και την περιφερειοποίηση των κανόνων εφόσον θα πρέπει να ενταχθεί το αίτημα του Κοινοβουλίου, δηλαδή η εφαρμογή της διαδικασίας συναπόφασης για τα βασικά στοιχεία της ρύθμισης και ο περιορισμός στις εξουδοτημένες πράξεις και επιτροπολογία για τις δράσεις που δεν είναι ουσιαστικές. Αυτά είχα να σας πω σχετικά με την έκθεση αυτή. κύριος Γκάλαχερ, παρακαλώ. Thanks, President. Just to thank... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για τη συνολική επισκόπηση του θέματος. Στην τελευταία μας συνάντηση ε, υπέδειξε ότι θα είχα κάποιο σχετικό πρόβλημα. Η συγγήτρια ανέφερε ότι παρατείνει το 2008 ο κανονισμός αυτός. Ξέρω ότι υπήρχαν τότε δυσκολίες και πέρασε το 2011. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον οι υπουργοί ε, αποφάσισαν κάτι στο Λουξεμβούργο πριν από την, ε, από την ε, εισαγωγή αυτής της ισχύω είχαν ελπίσει ότι θα είχαν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες πριν από τις 30 Ιουνίου του 2011. Βέβαια, υποστηρίζω την διατήρηση των μεταβατικών τεχνικών μέτρων και το έκανα επί σειρά ετών, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο τομέας αυτός και συγκεκριμένα τα αλληλευτικά αποθέματα θα μπορούσαν να αποφεληθούν. Το να επανέλθει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα και να ζητεί μια περαιτέρω παράταση 18 μηνών, εγώ σίγουρα δεν θα το υποστήριζα και θα το έθετα σαν τροπολογία. Το εναλλακτικό μου σχέδιο θα ήταν ε, να δώσουμε μια τέτοια παράταση μόνο εξαμήνου. Εγώ προέρχομαι από, από ένα δυτικό λιμένα της ε, Ιρλανδίας, όπου μικρά σκάφη κάτω από 15 μέτρα μπορούν να αλλιεύσουν μόνο στην παράκτια περιοχή. Αυτή η περιοχή και αναφέρομαι συγκεκριμένα και θεωρώ ότι αυτή η πολιτική είναι τοπική. Ε, σκέφτομαι συγκεκριμένα τις περιοχές ε, βορειοδυτικά της ε, Ιρλανδίας και βορειοδυτικά της Σκοτίας. Σημαίνει ότι οι μικρά σκάφη, τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκτυπο στα αλλιεύματα, δεν μπορούν να αλλιεύσουν στα νερά αυτά. Και όμως δεν είναι δυνατόν. Προφανώς και μπορούν να αλλιεύσουν. Ανάλογα μπορούν να... Τα 15 μέτρα σκάφη μπορούν να αλλιεύσουν ή μπορούν να πάνε προς νότον. Τα είδη τα οποία αλλιεύουν, κάποια αυτά δεν εμπίπτουν καν στις ποσοστώσεις άλλα είναι με ποσοστάσει, αλλά έχουν τόσο μικρά, τόσο, κάνουν τόσο, έχουν τόσο μικρές ψαριές, τόσο μικρά λιέματα που δεν έχει κανείς αντίκτυπο. Αντί να περιμένουμε λοιπόν την γενική αναθεώρηση κοινή αλληλευτική πολιτική, ελπίζω ότι θα είμαστε πολύ πιο λογικοί στα πλαίσια του εξωτολογισμού, όταν θα έχουμε αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο αναφέρεται, ε, σε τακτή βάση που αναφέρεται τις περιοχές ως οι παράκτιες νησιωτικές περιοχές. Ας το κάνουμε από τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Μιλάμε συνέχεια, αν θέλετε, για ε, επιμακρών, για μεγάλα σκάφη, για λιέμερα, για διάφορα ε, είδη. Αλλά εδώ δεν είναι πελασγικά τα είδη αυτά. Εμείς τους οθούμε τα μικρά αυτά σκάφη το πρέπει να πάνε, αν θέλετε, έξω στο πέλαγο για να μπορούν να έχουν κάποιε αντισταθμίσει. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι, είναι απειροελάχιστε οι ποσότητε οι οποίε αλλιεύουν και δεν έχουν καθένα αντίκτυπο. Τώρα έχουμε κάποια εξουσία μέσω τη συναπόφαση ω Επιτροπή Αλλία του Κοινοβουλίου. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Να συστήσουμε άμεσα τα μικρά αυτά σκάφη να μπορούν να αλλιεύουν στι μικρέ αυτέ περιοχέ. Βέβαια, δεν θέλω. Αν θέλετε, θα ξεκινήσουμε σε πιλωτικέ έρευνε. Δεν είναι μόνο η δική μου, αν θέλετε, αλλά και άλλε ε, αντίστοιχε μικρέ περιοχέ. Δεν υπάρχει καμία ποσόστοση ούτε του είδου ε, του αλλιεύματο και ούτω ή άλλω το ποσά, οι ποσότητε που αλλιεύουν δεν έχουν κανένα αντίκτυπο. Προφανώ είναι πολύ κοντά στην παράκτια περιοχή, αλλά ο στόχο θα πρέπει να είναι τα μεγαλύτερα σκάφη, τα οποία έχουν πραγματικό αντίκτυπο στα όλα αποθέματα. Θα ζητούσα λοιπόν από την Επιτροπή να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά να εισάγει ευελιξία για τα σκάφη που είναι μικρότερα από τα 15 μέτρα. Στο παρελθόν ήταν, ε, λεγόταν 50 πόδια. Και να, γίνει, να έχει άμεση ισχύ. Ή αν χρειαστεί κάποιος χρόνος για να παραταθεί ο κανονισμός αυτός, από την 1η Ιανουαρίου ή έστω από τις 30 Ιουνίου μέχρι το τέλος του χρόνου. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Αν είμαστε ρεαλιστές στην Επιτροπή, μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί να περιμένουμε μέχρι το 2013, όπως θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω η συγγήτρια να λάβει υπόψη την παρατήρησή μου αυτή. Θα πρέπει να ζητήσουμε και την Συμβουλευτική Επιτροπή από την περιοχή αυτή να μας πούν τι συμβαίνει. Εγώ ακούω τους αλείς στην ε, ακτές του Ντόνι Γκολ που ήμουν την περασμένη εβδομάδα με τον ε, Πρωθυπουργό το κύριο ανησυχία του ήταν εκεί, αυτή στην κύρια περιοχή. Η υγεία και ασφάλεια βέβαια είναι πολύ σημαντική, η και ασφάλεια στην τόπο εργασία του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι μπορεί να χρειάζεται να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να το κάνουμε εμεί εδώ στην Επιτροπή μα. Αν μη τι άλλο, αν θέλετε την εξασφάλιση υγιεινή και ασφάλεια και να δώσουμε σε αυτού του δυο τρει ανθρώπου, που αλλιεύουν στα μικρά σκάφη μια ευκαιρία να μπορέσουν να, ε, έχουν, να εξασφαλίσουν το επαστοζήν και να μπορούν να τις σταθμίσουν και να μην τους οθούμε έξω στο, στο πέλαγος. Γιατί πραγματικά, αν πέσουν και σε κακό καιρό, είναι πιθανότητα να ξεβραστούν στη ΣΥΠΑ παρά να επιστρέψουν στη Ιρλανδία. Προσωπικά, κύριε Γκάλαγκα, <clears throat> Νομίζω ότι αυτό το αίτημα, υπό το δικό μου πρίσμα προσωπικά θα έλεγα, είναι κάπως ε, επικίνδυνο, διότι διαφορετικά για κάθε ρακ θα έχουμε μια διαφορετική τοποθέτηση ως αίτημα ο ένας από τον άλλον. Και αυτό το οποίο ζητείτε αντί για παράταση θα είναι τροποποίηση του κανονισμού τεχνικών μέτρων. Και αυτό ακριβώς μετά την αποτυχία που υπήρξε όσον αφορά τα τεχνικά μέτρα με την πρόταση για κανονισμό στο παρελθόν που οδήγησε σε τροχοπέδηση, απόλυτη τροχοπέδηση από το Συμβούλιο. Αυτό που η Επιτροπή στοχεύει και η Επιτροπή μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα είναι στη μεταρρύθμιση να γίνει η ε, αναγκαία τροποποίηση και σε σχέση με το σύνολο της ε, αλληλευτικής πολιτικής και αυτό ακριβώς το 2013 που θα αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση να έχουμε τα τεχνικά μέτρα στη διάθεσή μας. Η Επιτροπή μπορεί να το, να το εξηγήσει καλύτερα. Εγώ απλά και μόνο λέω την προσωπική μου άποψη ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ ακαθόδες θέμα και να μην καταλήξουμε σε ανεπιθύμητες συζητήσεις τώρα εδώ γιατί για κάθε ράκο, όπως θα θυμόσαστε, Κάθε ρακ, για κάθε ρακ υπήρχαν πολύ διαφορετικές προτάσεις και πολύ θα έλεγα ε, συγκρουόμενες προτάσεις. Είναι επικίνδυνο αυτό. Δεν λέω ότι αν η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Αλληλείας ε, θέλει να κάνει αυτό που λέτε εσείς ε, δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Έχετε τον λόγο εσείς κύριε παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα από ότι εσάς θα πρέπει να αποφύγουμε να ανοίξουμε συζητήσεις ατελείωτες, ατέρμονες για μια πρόταση της Κομισιόν που έχει ως σκοπό μόνο να παρατείνει ένα υφιστάμενο σύστημα περιμένοντας να υπάρξει ένα νέο καθεστώς ε, για τα τεχνικά μέτρα διατήρησης μέσα στο πλαίσιο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Καταλαβαίνω ε, τα όσα είπε ο κύριος ε, Μάνελ Γκάλαγκερ, τις ανησυχίες του ε, και για τις εξαιρέσεις για μικρά πλοία. Καταλαβαίνω τις προτάσεις που έκαναν έξι άλλα κράτη-μέλη που μέσα στο Συμβούλιο έκαναν προτάσεις. Αλλά το θέμα που τίθεται είναι της λογικής μέσα στην μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής πρέπει να υποθεί. Η μεταρρύθμιση επειδή η παράταση αυτή θα επιτρέψει να υπάρξουν ορισμένα σημεία που θα συζητηθούν και που θα επαναπροσδιορίσουν την κατάσταση, ενώ αυτό πρέπει, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει νέο πλαίσιο. Η Κομισιόν πιστεύει ότι όχι και δέχεται να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα, αλλά μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο διαφορετικό, το πλαίσιο της μεταρρύθμισης. Γι' αυτό το θέμα του κυρίου Γκάλαβέρ για τα μικρότερα πρία κάτω από 112 κιλοβάτ που είναι ε, στα νυχτά της Σκοτίας θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο μεταρρύθμισης της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και όχι παράτασης αυτού του νομικού καθεστώτος. Ευχαριστούμε ε, την εισηγήτρια που ακολουθεί την λογική της Επιτροπής και προτείνουμε συνεπώς να δόθει συνέχεια στην έκθεση αυτή με μια παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 αυτού του μηχανισμού και τότε θα πρέπει να έχουμε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης ένα νέο μηχανισμό ε, για τα ε, τεχνικά μέτρα διατήρησης. Έχουμε την αιτιολογική έκθεση της εισηγήτριας και βεβαίως θα ακολουθήσουμε Επιμελώσα, θα παρακολουθήσουμε τις αρμοδιότητες ε, του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτά τα ουσιαστικά και μη ουσιαστικά ε, στιμία ε, που αποτελούν στοιχεία κατετοξιοδότηση πράξεων. Ευχαριστώ. Να διευκρινίσω κάτι στην Ευρω... στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι είμαστε στην ίδια θέση. Το γεγονό ότι δεν προβλέπουμε και προκαταλαμβάνουμε την μελλοντική κοινή αλληλευτική πολιτική. Ναι, παρόλα αυτά που συμφωνούμε, τον Ιούνιο του 2011 μέχρι άλλου 18 μήνες παράτασης ισχύω κανονισμού να αποτελέσουν αντικείμενο, αν θέλετε, αξιολόγηση αυτών των περίφημων τεχνικών μέτρων. Θέλω να σα ε, διασφαλίσω ότι θα παραμείνει αυτή η αξιολόγηση και δεν υπονοείται, αν θέλετε, σαν κάποια νέα ΚΑΠ. Θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε αυτό το σημείο. Το εννοούμε έτσι. Uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι είναι κινδυνευμένο, αλλά μόνο όταν μιλάμε για τον κίνδυνο να οθούμε τα μικρά σκάφη στα νυχτά του Ατλαντικού. Όχι επικίνδυνο έτσι όπως συμφωνήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως το είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απογοητεύομαι, είμαστε εδώ για να ακούσουμε την θέση όλων των μελών και εσείς πρέπει να προεδρεύετε όλων αυτών των απόψεων. Εάν πρόκειται να είναι, αν θέλετε, κλειστό το θέμα, δεν θα μιλούσαμε για κάτι προηγούμενο. Θα πρέπει να είμαστε έντιμοι και ανοιχτοί στην Επιτροπή αυτή. Έχει πριν από πάρα πολύ καιρό ξαναθύμωσα, αλλά ξανά είμαι θυμωμένο τώρα. Α είμαστε πραγματιστέ. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι ακριβώ υπάρχει αυτή η Επιτροπή. Θα πρέπει να έχουμε αδιαμαρτύρητα την θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν άλλε εκθέσει που δεν αποδέχονται αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λέω. Α εξετάσουμε τη συνείδησή μα, α το σκεφτούμε τι επόμενε εβδομάδε Ας ασκήσουμε κάποια πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τους δώσουμε ένα εξάμεινο και εν τω μεταξύ θα πρέπει να έχει πληχθεί κάποια ευελιξία και κάποιες παρεκκλήσεις. Και εγώ μιλάω αν θέλετε από θέση, αν θέλετε αυθεντίες, γιατί εκπροσωπώ μία από τις χώρες εκείνες που έχουν που δεν μπορώ να το πω άμεσα, θα το πω όμως έμεσα. Υπάρχουν κάποιε χώρε οι οποίε ξεπερνούν κατά πολύ τι ποσοστώσεις, κατά εκατοντάδε. χιλιάδες τόνους. Και θα την κατονομάσω τις χώρες αυτές στο άμεσο μέλλον, θα έχω την ευκαιρία. Α δούμε λοιπόν τα μεγάλα σκάφη που το κάνουν αυτό. Γιατί εμεί στην Ιρλανδία έχουμε κάνει καταγγελία. Υπάρχει έλεγχο, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο των υπολείπων χωρών, όπου παίρνουν εκατοντάδε. χιλιάδες ε, τόνους ε, αλλιευμάτων στην κυρίω Ευρώπη. Εγώ, κύριε Γκάλαχερ, και εγώ μπορώ να εκφράζω την άποψή μου. Έχω την, την προσωπική μου άποψη. Γι' αυτό είπα ότι αν συμφωνούν η πλειοψηφία των μελών να κάνουν κάτι άλλο, εντάξει. Αλλά εγώ είμαι ευρωβουλευτή, να είμαι πρόεδρο και έδωσα την προσωπική μου άποψη. Μπορεί να είναι σφαλμένη η άποψή μου, αλλά είναι η άποψή μου αυτή. Και έχω και εγώ δικαίωμα να εκφράζομαι, έτσι. Δεν έχω παρά και τη δική μου άποψη. Και αυτήν εκφράζει ο καθένα. Είπα ότι αν η πλειοψηφία θέλει να κάνει κάτι άλλο, εντάξει, να ανοίξει η διαδικασία. Καμία αντίρρηση. Εγώ έδωσα τη δική μου άποψη και υπό τη δική μου άποψη δικαιολογούνται οι λόγοι που με έκαναν να πω αυτά τα οποία είπα. Κύριε Κυρία Πρόεδρε, ήθελα καταρχάς να απαντήσω στην εισηγήτρια στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν στοχεύει, αν θέλετε, να κοφεύσει στις προτάσεις που τις γίνονται, κάθε άλλο. Και μάλιστα αποδεικνύεται ότι οι προτάσεις οι οποίες υπευλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο, ιδιαίτερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελούν αντικείμενο ε, αξιολόγησης από την SSTF και θα υπάρχουν προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν και την πιθανότητα παρεκκλήσεων και την χρήση διαφορετικών μηχανισμών σε σχέση με τα διαφορετικά σκάφη και τις ε, μηχανές μέχρι 1112 κιλοβάτ, όπως αναφέρει ο κύριος ε, Γκάλαχερ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την νομοθετική έκφραση στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, δεν θέλουμε να παρατείνουμε με τα υφιστάμενα μεταβατικά τεχνικά μέτρα, γιατί τα χρειαζόμαστε πέραν της 30 Ιουνίου του 2011. Γιατί, Γιατί οι αξιολογήσει αντίκτυπου που πραγματικά μας επικρίνονται ότι δεν είχαμε κάνει πέρσι τον Νοέμβριο, όταν παρουσιάσαμε τα μέτρα, τα τεχνικά μέτρα, τις κάνουμε σήμερα, έχουμε δεσμευτεί να το κάνουμε. Αυτές οι αξιολογήσεις ε, περιβαλλοντικού αντίκτυπου απαιτούν χρόνο, δυστυχώ έτσι έχουν τα πράγματα. Μελετάμε λοιπόν τα αιτήματα αυτά πολύ σοβαρά, Έχουμε αυτή τη στιγμή μισή ντουζίνα, αν θέλετε, σχεδίων αυτών. Τώρα σκεφτόμαστε την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ακριβώς μετά από αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου και ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να υποβάλουμε κάτι στα πλαίσια ακριβώς και μετά από το πέρας αυτής της περίοδου ε, παράτασης του υφιστάμενου καθεστώτος και επί τη βάση των προτάσεων που έχουν γίνει. Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα παρεμβεσίτης. Καθορίζουμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα που ελπίζω ότι θα συμφωνείτε κυρία Συγχύτρια η κατάθεση τροπολογιών. 15 Δεκεμβρίου το μεσημέρι ψήφιση στην Επιτροπή 25-26 Ιανουαρίου ψήφιση στην Ολομέλεια. Καταρχήν ε, την ε, επόμενη Ολομέλεια. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε με το 7 και περνάμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα πριν περάσουμε στη συνάντηση των συντονιστών που είναι το 9. Συμφωνία, συμφωνία αλληλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μικρονησία. Εγώ είμαι η για αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρώτα τη δική της, το δικό της σχέδιο. Έχετε κύριε Μιλά τον λόγο παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στην αγγλική καμπίνα ότι το όνομά μου είναι Αμιάπ. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω αγγλικά για να πω ότι αυτός ο τομέας, αυτή η ζώνα, η ζώνη είναι η πλουσιότερη ε, για τον, την αλία Αθηνοειδών. Υπάρχουν πάρα πολλά αποθέματα ακόμα. Ε, μερικά βρίσκονται υποποίηση, παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δυτικό Ειρηνικό είναι μέτρια σε σχέση με την παρουσία ανατολικά όπου παραδοσιακά η, ο στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δραστηριοποιείται κυρίως επειδή υπάρχουν πολλές επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λατινική Αμερική και βεβαίως εκφορτώνουν στις χώρες αυτές πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως αυξανόμενο ενδιαφέρον ε, ο στόλος ε, αλίας θηνοειδών να δραστηριοποιηθεί δυτικά. Ο ένας λόγος είναι επειδή υπάρχουν ε, δυνατότητες αλλιευτικέ σημαντικές όπως είπα, αλλά και κυρίως επειδή όπως είπαμε προηγουμένως υπάρχει ανάγκη για το στόλο μας να βρει ε, νέες ζώνες αλίας. Έχουμε ε, τρεις συμφωνίες στον Ειρηνικό, με Κυριμπάτη, με τα νησιά Σολομόντος. Αυτή η συμφωνία συζητείται σήμερα ε, με τις Ομοσπονδιακές Πολιτείες της Μικρονησίας διαπραγματευόμαστε, την διαπραγματευτήκαμε το 2004 τη συμφωνία και τέθηκε σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2007 με το πρώτο πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο που συζητείται σήμερα για ενδεχόμενη ανανέωση για τρία χρόνια από το 2007 μέχρι το 2010. Το πρωτόκολλο αυτό δεν υλοποιήθηκε πραγματικά παρόλο που τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι εφοπλιστές είχαν πληρώσει την συνδρομή τους, τη συνεισφορά τους στη Μικρονησία για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με τις δυσκολίες κυρίως πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα που θα μπορούσε να λειτουργήσει κανονικά. Έγιναν όμως αυτές οι καταβολές, αλλά δεν δόθηκαν άδειε από τη Μικρονησία σε πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσεις συνεχίζονται και το πρόβλημα των πληρωμών, των καταβολών αυτών που έγιναν, αλλά δεν ε, είχαν κανένα αντίκρισμα, συζητήθηκαν με τους εκπροσώπους της Μικρονησίας. Το νέο πρωτόκολλο μονογραφήθηκε τον Μάιο του 2010. Η διάρκεια του πρωτοκόλλου θα πρέπει να είναι πενταετής και αυτό ε, συμπίπτει με την υπολείπουσα ε, διάρκεια υλοποίησης της ίδιας της συμφωνίας. Όπως και στην προηγούμενη συμφωνία με τις Κομόρες οι τόνοι αναφερόμενοι έχουν μειωθεί ε, σύμφωνα με τις υποστημονικές συμβουλίες διότι στο μείγμα ε, των ειδών που αλλιεύονται ε, έχουμε μερικά είδη τα οποία δεν έχουν τόσα αποθέματα. Μπορεί ο κίτρινόπτερος τόνος να έχει αποθέματα, αλλά άλλα δεν έχουν αποθέματα. Θα έπρεπε ε, λοιπόν να υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες, υπάρχουν ε, έξι πλοία ε, γρηγροί, έξι παραγαδιάρι, πέντε παραγαδιάρικα που ενδιαφέρονται. Υπάρχουν συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, υπάρχουν πλοία περιπολίας και πλοία με άλλες, με ε, θα παραμείνει ίδια η ε, συνεισφορά, αλλά για τους ίδιους λόγους όπως για τις ε, κομόρες η πρόσβαση θα αντισταθμιστεί με μια αύξηση του τμήματος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για υποστήριξη της τομεακής πολιτικής στην Μικρονησία. Επίσης συμφωνήθηκε ότι θα ρυθμιστεί το χρέος της Μικρονησίας με μείωση τόσο του ποσού που θα καταβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον προϋπολογισμό της χώρας, αλλά και αντιστάθμιστη για τα ποσά που καταβλήθηκαν προηγουμένως από τους εφοπλιστές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την πρώτη περίοδο της συμφωνίας και ότι τώρα οι άδειε θα πρέπει να δοθούν δωρεάν και ότι δεν θα γίνουν άλλες καταβολές και πληρωμές για το, την δεύτερη περίοδο. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα αυτή είναι η θέση στην περιοχή και το γεγονός ότι ως μέλος της WFCPSC που είναι η Επιτροπή Αλίας ε, Κεντρικού και Δυτικού Ειρηνικού, η οργάνωση η οποία θέτει τους ε, κανόνες ε, για την περιοχή, το πρωτόκολλο, το διμερές το οποίο υπογράφουμε με την χώρα αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα μέτρα ε, τα οποία έχουν υιοθετηθεί για να ρυθμιστεί η αλίευση θηνοειδών στην περιοχή. Θα πρέπει οι ξένες χώρες να λάβουν υπόψη ότι η WFCFP ε, θα πρέπει να παρακολουθεί, να επιτηρεί. Υπάρχει ένας παρτηρητής σε όλα τα πλοία γρηγρή τα οποία αλλιεύουν ε, στις περιοχές αυτές. Επίσης, στην συμφωνία προβλέπεται ότι θα υπάρξει ένας ναυτικός ε, του τόπου ε, σε κάθε πλοίο. Νέες ρήτρες έχουν εισηχθεί στην ε, συμφωνία αυτή όπως ανέφερα και για την προηγούμενη περίπτωση, θα είμαι σύντομος μια διάταξη αποκλειστικότητας για τα πλοία, μια ρήτρα αναθεώρησης για τροποποίηση του πρωτοκόλου σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής στις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής. Πίσω από αυτή τη φράση υπάρχει αναφορά στην μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής κυρίως και στις συμφωνίες συνεργασίας αλλιευτικής και επίσης διαρρήτρα διακοπής, αναστολής σε περίπτωση παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή αναστολής της συνεισφοράς της οικονομικής αν τα όσα συμφωνήσαμε με τη χώρα για την ανάπτυξη της αλλιευτικής πολιτικής δεν έχουν τηρηθεί. Εκεί βρισκόμαστε τώρα, αυτή είναι η κατάσταση. Εξετάζουμε την κατάσταση και περιμένουμε τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το νέο πρωτόκολλο. Από τη δική τους πλευρά οι αρχές της Μικρονησίας έχουν εξετάσει το πρωτόκολλο αυτό ενδελεχώς και έχουν περάσει στην διαδικασία επικύρωσης και ελπίζουμε ότι τον Ιανουάριο θα γίνει η επικύρωση τον Ιανουάριο του 2011. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Eh, Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Αμιάτα. Κυρία Αμιάτα. Πολύ καλά συνοψίστηκε το θέμα της μικρονησίας από πλευρά. Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι συνάδελφοι αυτό που αναφέρθηκε ότι υπάρχουν τρεις συμφωνίες αλίας, νήσος Σολομόντος, Κυριμπάτη και της Μικρονησίας. Και η σημασία που έχουν αυτές οι τρεις συμφωνίες αλίας με χώρες που είναι χώρες ΑΚΕ. Η Μικρονησία εντάχθηκε στις ΑΚΕ το 2000 ε, ε, και έχουμε και την συμφωνία της ΛΟΜΕ και έχουμε και την συμφωνία για την ανάπτυξη και τη συνεργασία για την ανάπτυξη με όλη αυτή τη ζώνα. Έχουμε λοιπόν μεγαλύτερο εύρος από ότι αποκλειστικά την Αλία. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε οι συνάδελφοι επίσης ότι πέρα από την τοπική οργάνωση αλίας που είναι η Western Pacific Fisheries Commission του Δυτικού Ειρηνικού δηλαδή Επιτροπή Αλίας. Έχουμε και τη Συμφωνία Παλάου, του Παλάου και τη Συμφωνία του Ναούρου που είναι δύο συμφωνίες ε, υποπεριφερειακές που και αυτές εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπό άλλη αιγίδα του δυτικού ε, ειρηνικού, υπό άλλη στέγαση θα έλεγα, άλλη ομπρέλα. Λοιπόν, για αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς που πολύ σωστά αναφέρατε κύριε Αμιάτη είναι οι πιο πλούσιες ε, οι νήσοι αυτές της Μικρονησίας ε, σε θηνοειδή, σε τονοειδή. Μεγάλο ποσοστό των ε, παγκοσμίων αλλιευμάτων προέρχονται από εκεί, του, δι, του δυτικού ειρηνικού. 80% είναι πολύ πλούσια σε αλλιεύματα νερά αυτά. Μια υδάτινη περιοχή πάρα πολύ χρήσιμη. Η Ευρωπαϊ, ο Ευρωπαϊκός Στόλος έχει 7 μεταξύ 6 και 7 ε, παραγαδιάρικων και ε, ένα αντίστοιχο αριθμό γρηγρή είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτός ο στόλος εκεί και γι' αυτό αυτές οι συμφωνίες για αυτή τη ζώνη νήσου Σολομόντα, Κυριμπάτη και Μικρονησία είναι λοιπόν μια ε, καλή δουλειά όσον αφορά την περιοχή, την υποπεριφέρεια αυτή όπου επιπλέον έχουμε και τα θέματα προστασίας ε, και του Western Pacific και του Παλάου και Ναούρου. Η ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών των θεμάτων και της ε, χρήσης ε, των, για τα αλλιεύματα αυτά και κάτι το αξιοπερίεργο που φαίνεται ότι οι πληρωμές θα γίνονται λέει σε ευρώ και η Μικρονησία είχε ένα λογαριασμό μόνο σε δολάρια και αυτό δημιουργεί κάποια αξιοπερίεργα θέματα. Χρόνια θα πάρει να επιληθεί αυτό. Αυτό ε, για τις προσοχής μου, διότι σε σχέση με τα, τα συνομόσπονδα κράτη της ε, Μικρονησίας να έχουν ένα λογαριασμό, λέει, σε ευρώ και να πρέπει να καταβάλλονται αυτά τα ποσά σε ευρώ και όχι ε, στο δικό σου λογαριασμό. Αυτό έχει γίνει πρόβλημα κρατικό θα έλεγα, το οποίο δυσκολεύει την εφαρμογή της συμφωνίας. Κυρίως όπως, όταν είπατε εσείς έχουμε και την ε, αντιστάθμιση, την καταβολή της χρηματικής αντιστάθμισης και όπως είπατε οι εφοπλιστές πλήρωσαν. Από ό,τι γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, η συνέχεια λέγεται για τέσσερις, ε, για τις άδειες τεσσάρων για, αυτό θα σήμαινε ε, συν επιπλέον για τους παρατηρητές, συν την αδειοδότηση, οι εφοπλιστές ε, πλήρωσαν αλλά δεν μπόρεσαν, δεν μπορούν να αλλιεύσουν. Τι γίνεται με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μας το επεξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί από το 2007 όλα αυτά δεν έχουν, ε, ας το πω έτσι, επιληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω απόλυτα. Υπάρχει υποχρέωση σε αυτή τη ζώνη όλοι οι τομεί να έχουν ένα παρατηρητή, όλα τα σκάφη να έχουν ένα ε, παρατηρητή. Παραγαδιάρικα, γρηγρή κτλ. Προφανώς πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Αν όμως διαβάσει κανείς τη συμφωνία, τι βλέπει. Και παραγαδιάρικα και γρηγρή, από ό,τι βλέπουμε εδώ, για να έχουν την άδεια, πρέπει να πληρώσουν ποσοστά ποσά για τον παρατηρητή επιπλέον. Αυτό συμβαίνει. Εγώ τουλάχιστον αυτό αποκόμισα από την ανάγνωση του πρωτοκόλου. Πέρα από την αδειοδότηση, γρηγρή και παραγαδιάρικα να πληρώνουν επιπλέον το ποσό για έναν επόπτη, για έναν παρατηρητή. Ερωτώ, σωστή η ερμηνεία μου αυτή ή όχι. Διότι αν έχουμε λοιπόν και κάλυψη κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό όπως είναι υποχρεωτική, τι γίνεται με τα γρηγρή και τα παραγαδιάρκα, σε τι οφείλεται αυτή η κατάσταση. Υπάρχει μετά ένα τρίτο στοιχείο που είναι και αυτό σημαντικό. Και αυτό είναι ότι στην έκθεση αξιολόγησης γιατί πριν από την τελευταία αυτή απόφαση που είχαμε, είχαμε αυτά τα στοιχεία, λέει αυτή η έκθεση αξιολόγησης κάτι ενδιαφέρον, μου φαίνεται. Τώρα έχοντας αυτές τις συμφωνίες για αυτή τη ζώνη και επιπλέον εμένω και επιμένω μέσα στην πολιτική μια στρατηγική συνεργασίας ευρύτερου πλαισίου, ευρύτερης εμβέλειας όπως αυτή που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το European Development Fund, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, έτσι, τα σχετικά κονδύλια για την ανάπτυξη ε, αυτών των περιοχών. Διαρωτώ με, σε σχέση με την έκθεση αξιολόγησης, δεν θα ήταν σκόπιμο να υπήρχε μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να πάει σε αυτή τη ζώνη και να επιτηρήσει τι γίνεται, να υποπτεύσει την κατάσταση. Τώρα, από το 2006-2007 θα μπορούσε να, να είχε επιληθεί το θέμα των προκαταβολών και των πληρωμών. Παρ' όλα αυτά, καλό θα ήταν ε, δεδομένων αυτών των προβλημάτων να υπάρχει παρατηρητήριο εκεί, μια αντιπροσωπεία σε αυτή τη ζώνα. Σε αυτή τη ζώνα ξεκινά μια ανάπτυξη αλλιευτικών δραστηριοτήτων. Γιατί λοιπόν και, χτίζονται αυτές οι δραστηριότητες ε, ευθύ εξ αρχή, γιατί δεν αποστέλει, δεν έχει μια αντιπροσωπεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί και όπως είπε ο κύριος ε, Καπόλας, και εγώ θα το προτείνω στην έκθεσή μου, όπως εκείνος θα προτείνει κάτι αντίστοιχο, να υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί, να μπορεί να επιτηρήσει και να ελέγξει κάπως τα πράγματα για τα όσα γίνονται εκεί. Τι λέτε. Να, μας πληροφορεί, να, να έχουμε πληροφορίες σχετικά και για την Παππούα Νέα Γουινέα που είναι τόσο κοντά εκεί. Τέλος πάντων, έστω να έχουμε πληροφόρηση από πρώτο χέρι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέτω έτσι. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Θα ήθελα επ' αυτόν και σε σχέση και με την, ε, ε, το εύρωστο των αλλιευτικών δραστηριοτήτων όπως με το τονάς που αναφέρεται. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και με το ξυφοειδές, τέσσερα ή έξι ε, παραγαδιάρικα ασχολούνται με αυτό, αλλά η Επιστημονική Επιτροπή για την Αλία πρότεινε μείωση μείωση των αλληλευτικών δραστηριοτήτων για το ξυφοειδές. Και εδώ έχουμε πολλά στοιχεία ε, σε σχέση με το πρωτόκολλο. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτές τις ερώτησεις. Η κυρία Άντρες Μπαρέα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς καταρχήν θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συμφωνία, διότι πρέπει να συνεχιστεί ο στόχος της ανάπτυξης, της συνδρομής και υποστήριξης του τομέα και του ανεφοδιασμού των αγορών και για την ευρωπαϊκή παρουσία στη ζώνη που είναι σημαντική. Διότι έχουμε εδώ και την άσκηση των αλλιευτικών αυτών δραστηριοτήτων και για την ανάπτυξη της ζώνης αυτής και μέσω της βοήθειας για την ανάπτυξη αυτό το αρχιπέλαγος των 605 μικρών νήσων πρέπει να υποφεληθεί, να βοηθηθεί από μας. Εσείς ε, αναφερθήκατε σε σχέση με τις πληρωμές, ε, ε, είπατε ότι υπάρχουν ελλείψεις και υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να επιληθούν αυτά, δεν είναι πρόβλημα ενός λογαριασμού μόνο. Πρέπει να τεθεί εντάξει να μπουν στα σωστά πλαίσια αυτά για να μην υπάρχουν προβλήματα και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να επιλύει αυτά τα προβλήματα χωρίς να υπάρχουν ζημιές, ε, να υπάρχει επιβάρυνση ούτε για τη Μικρονησία ούτε για τον τομέα τον αλλιευτικό που δραστηριοποιείται από εμά από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Επίσης για τη δυνατότητα να υπάρχει ένα παρατηρητήριο εκεί ή μια αποστολή παρατηρητών όπως είπε η Πρόεδρος για να αξιολογηθούν οι συμφωνίες αυτές και τι γίνεται με αυτές και να είναι πραγματιστική προσγειωμένη η προσέγγιση μας να δούμε τι γίνεται από πρώτο χέρι, να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση σε σχέση με αυτά. Οι δυο μας λοιπόν συμφωνούμε. Πάντα συμφωνούμε όταν θέλουμε να βελτιωθούν τα πράγματα σε σχέση με ελλείψεις και να προβλήματα που υπάρχουν και πρέπει να εξηγιανθούν και να τεθούν εντάξει. Και φυσικά για την ε, μικρονησία και ε, να ε, μπορούμε από εκεί να δράσουμε και για την Παππούα είναι Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την παρουσίαση της κατάστασης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσέγγιση που θέλει να δει η Επιτροπή με πολύ πιο φιλόδοξο τρόπο και σε περιφερειακό επίπεδο τη συμφωνία αυτής, καθώς και τη διαχείριση των αλλιευτικών πόρων. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στην εκμετάλλευση των πόρων ναι. αυτών. Είναι μια καλή προσέγγιση λοιπόν. Εξακολουθώ όμω να είμαι λίγο προβληματισμένη. Σε κάθε μία από αυτές τις αξιολογήσεις των συμφωνιών που μελέτησε, είδα ότι στα συμπεράσματα, η γενική, αν θέλετε τα συμπεράσματα καταρχάς, είναι ότι καμία από αυτές τις συμφωνίες δεν έχει πληρώσει τους στόχους της. Και αυτή είναι ουσιαστικά η αρχική φράση του συμπεράσματος κάθε αξιολόγησης, ότι έχει υπολείπεται των συνολικών στόχων που έθεσε η συμφωνία. Και οι συστάσεις οι οποίες ακολουθούν σε κάθε συμφωνία και τη συμφωνία με τα νησιά του Σολομόντος και στην λόγο Συμφωνία και στις Κομόρες, είναι ότι η σύσταση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδικό προσωπικό το οποίο θα εγκατασταθεί στην περιοχή. Και κάθε εφαρμογή, αν υπάρχει κάποια εφαρμογή στις χώρες αυτές, θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, ηγούμενος εταίρος, αν θέλετε, και θα πρέπει να πρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται μάλιστα ότι η διαχείριση αυτών των συμφωνιών ε, του ειρηνικού από τα κεντρικά γραφεία των Βρυξελών δεν είναι λύση και είναι πολύ κέρια η παρατήρηση αυτή. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ακριβώς όπως η κυρία Πρόεδρος, κατά πόσο αν υπάρχουν συγκεκριμένες ιδέες στο να εγκατασταθεί προσωπικό στην περιοχή εκεί, ώστε αυτές οι συμφωνίες να είναι πραγματικά εταιρικέ ε, συμφωνίε, εταιρικέ σχέσει. Είναι πραγματικά γελίο να ακούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε σε αυτή την περιοχή. Χρειάζονται πέντε μέρε ταξίδι. Μα πληρώνουμε για αλληλευτικές ευκαιρίες για τους ευρωπαϊκούς αλληλευτικούς θόλους να πάνε εκεί και επομένως έχουμε την αντίστοιχη ευθύνη να εξασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες αυτές θα εφαρμόζονται σωστά και υπεύθυνα. Και αυτό με οδηγεί στην δεύτερη παρατηρήσή μου, σχετικά με την κατάσταση των αλλιευμάτων. Στην έκθεση αξιολόγησης διαβάζω ότι ο κυτρινόπτερος ε, τόνος είναι μόνο 30% των λιμμάτων και υπάρχει υπεραλίευση των, ε, των άλλων ειδών τόνου και ότι τα στοιχεία για τον πληθυσμό των καρχαριών δεν είναι καθόλου αξιόπιστα. Έχουμε όμως με τις σχετικές συμφωνίες αλίες και την αρχή ότι δεν θα εκμεταλλευόμαστε, δεν θα υπερεκμετάλλευση κανενός αλλιεύματος, κανενός είδους, επουδενή και σίγουρα κανένα λίμα που θα μπορούσε να είναι προ όφελο του ντόπιου πληθυσμού. Σε αυτή την περίπτωση όμω, πληρώνουμε μόνο για πρόσβαση συγκεκριμένου αριθμού σκαφών και το να μην θέτουμε αρκετές ποσοστώσεις για κανένα είδος. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε πραγματικά ότι δεν συνεισφέρουμε και εμείς στην ε, υπερα, υπεραλίευση της, ε, του κυτρινόπτερου ή του ερυθρόπτερου ε, τόνου ή του Άρα πώς ξέρουμε πώς μπορούμε Αυτά τα σκάφη μπορούν να λιεύσουν οτιδήποτε, ακόμα και καρχαρίες ε, ή, ή θαλάσσια πτηνά ή και χελώνες. Άρα πώς ξέρουμε, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τι ακριβώς αλλιεύουν τα σκάφη αυτά φτάνοντας εκεί. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ε, Κυρία Μπιλμπάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις εξηγήσει που έδωσε. Καταρχήν είμαι υπέρ του να έχουμε συμφωνίες αλίας που όπως ακριβώς αναφέρθηκε δεν θα περιορίζονται μόνο στη Μικρονησία, αλλά θα πρέπει να δούμε τις τρεις συμφωνίες αλίας συνολικά, σφαιρικά για τον ειρηνικό, το δυτικό ειρηνικό με τα νησιά Σολομόντα, Κυριμπάτη και Μικρονησία. Είμαι υπέρ λοιπόν διότι είναι υποφελή για τον τομέα μα, τον τομέα τη Αλία. Και να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση ότι συμφωνώ με τι νέε ρήτρε που εισήχθησαν σε αυτή τη συμφωνία και που κάνουν λόγο για την αναθεώρηση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την παραβία, σε περίπτωση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και το τι θα γίνει σε περίπτωση μη τήρησης όλων αυτών. Αυτά τα μέτρα ελέγχου ενισχύουν πιστεύω. Θα έπρεπε να μπορούν να βοηθήσουν να ενισχύσουν την εικόνα του στόλου και των ε, αλευτικών δραστηριοτήτων. Εμένω και επιμένω. Είναι μια ανησυχία αυτή. Ένα μέρη, μια μέρημνα που όχι μόνο έχω εγώ αλλά και όλο ο τομέα αλίας. Όλο αυτό το περιεχόμενο με όλες τις νέες αυτές διατάξεις να βοηθήσει, να μπορέσει να βοηθήσει να δοθεί μια διαφορετική εικόνα από αυτή που δίνεται από τον τομέα της αλληλείας ε, σήμερα. Ως προς αυτό θα πρότεινα να γίνει κάποια προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να αναγνωριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό, τους, υπό τις και τους οποίους ε, δρά ο αλληλευτικός στόλος. Αυτό σε σχέση με τις αλληλευτικές δραστηριότητες, διότι οι επιστημονικές εκθέσεις αυτό προτείνουν σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές και να αναμείνουμε να δούμε, να ελπίσουμε ότι η συμφωνία αυτή θα έχει την υποστήριξη των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υποστήριζα την πρόταση της Προέδρου εγώ. Είναι μια καλή πρόταση θα έλεγα. Πρόταση για να βελτιωθεί η λειτουργία, η λειτουργία των συμφωνιών αυτών θα έπρεπε να πούμε ότι είναι υπερβολικό το διάστημα το οποίο διαρκεί αυτό το θέμα. Τρία χρόνια για την μεταφορά κονδυλίων, για την εξόφληση ποσών. Θα έπρεπε λοιπόν ήδη το πρώτο έτος να έχουμε ρύθμιση των θεμάτων αδειοδότησης αδειών αλίας. Θα έλεγα λοιπόν με αυτό το περιεχόμενο να βελτιωθεί η εικόνα τη Αλία. Θα πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ειδική ξεχωριστή προσπάθεια για να προχωρήσουν όλα αυτά. Και έχουμε μια διοικητική πρόταση υποστήριξης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ευχαριστώ. Ε, Θα πάρω με τη σειρά τα ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά την ε, αποζημίωση των ε, πλειοκτητών, Επαναλαμβάνω ότι συμφωνήθηκε με την ε, Μικρονησία ότι η έκδοση αδειών αλλιεύσης κατά διάρκεια του πρώτου έτους ισχύω του νέου πρωτοκόλου θα γίνεται δωρεάν, χωρίς επιπρόσθετη καταβολή κάποιας ε, ε, αμοιβή σε αντιστάθμιση, αν θέλετε, των χρημάτων που δαπανήθηκαν στα προηγούμενα χρόνια και που δεν οδήγησαν τελικά στην παράδοση σχετικά έκδοση σχετικών αλλιευτικών αδειών. Έτσι λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει αναχρηματοδότηση, αν θέλετε, του χρέου αυτού. Το χρέο που αφορά και την πληρωμή που καταβλήθηκε από τον κοινωνικό, κοινοτικό προπολογισμό θα αντισταθμιστεί ε, ε αφαιρώντα ε, τα ετήσια ποσά σε σχέση με τη συνολική εισφορά που θα καταβληθεί στην Μικρονησία. Θα ήθελα να πω και λίγα λόγια σχετικά με την σύνδεση ε, μεταξύ της αναπτυξιακής αρρωγής και της ε, εταιρική σχέσης αλίας των σχετικών συμφωνίων που έχουν υπογραφεί. Είναι αλήθεια ότι μεγάλα ποσά δαπανήθηκαν στην περιοχή, ιδιαίτερα για να βοηθηθεί η επιστήμη. Από το Αναπτυξιακό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Να πούμε ότι, ότι αυτό έγινε σε πλήρη συντονισμό με την Γενική Διεύθυνση Αλίας ε, ή ε, τις προηγούμενες τις προκατόχους ε, διευθύνσεις. Θα ήταν πραγματικά υπερβολή μόνο συντονισμό δεν υπήρξε, αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρήματα αυτά συνεισέφεραν τα μάλα στην βελτίωση του επέδου τεχνογνωσία και επιστήμη στην περιοχή. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα για να υπάρξει συνοχή και συνέχεια μεταξύ των εταιρικών ε, σχέσεων ε, αλληλεία, τη συμφωνία ε, εταιρική σχέση, αλληλευτική σύμπραξη, των συμφωνιών αλληλευτική σύμπραξη και του Αναπτυξιακού Ταμείου. Το σημαντικό που πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι η αλλιευτική σύμπραξη εν γέννη γίνεται και οι δαπάνες και εκταμιεύσεις γίνονται από πολύ σαφείς και αυστηρούς ε, ε, κύκλους προγραμματισμού που είναι συνήθως μακρύς, 5-6 ετών και που βασίζονται σε μια πάρα πολύ βασική αρχή. Και αυτή η αρχή είναι ότι θα πρέπει να συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό τομέων. Και αυτή είναι και η επιλογή των χωρών που ε, είναι δικαιούχοι και υποφελούνται από την αρρωγή αυτή. Πολύ σπάνια υπάρχει ε, από τους δικαιούχους συγκέντρωση των αλλιευτικών τομέων, συγκέντρωση ένα τομέα. Μπορούμε σαφέστατα να βελτιώσουμε την όλη συνοχή της προσέγγισης, αλλά σίγουρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές, τις διαφορετικές μεθοδολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ε, δαπάνη και την εφαρμογή αυτής της ε, αρρωγής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην περιοχή, πολύ σωστά αναφέρατε κυρία Πρόεδρε, ότι καταρχάς υπάρχει ένα πολύ ψηλό επίπεδο περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών στην ε, περιοχή εκείνη. Μας προβληματίζουν όμως κάποιες πτυχές αυτής της περιφερειακής συνεργασίας. Η όλη συμφωνία για τα επικαλυπτόμενα αλλιεύματα, ε, όπως η σχετική συμφωνία για την ε, δυτικό ειρηνικό βασίζεται, ε, βασίζεται σε αυτή την γενική αρχή πρόσβασης στα λιεύματα. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν σε αυτήν την ε, στενή τη ενία συμφωνία που αναφέρουμε είναι ότι οι χώρες αυτές προσπαθούν να κλείσουν την πρόσβαση στις, ε, στην πελαζική αλία, ώστε η αλία να γίνεται εντός χωρικών υδάτων εμποδίζοντας ουσιαστικά τους τόλους να έχουν ε, ελεύθερη πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα και εμποδίζοντας επίσης και τον φορέα ε, του Δυτικού Ειρηνικού ε, και της Συμφωνίας WPFC να διδραματίσει το ρόλο του ω φορέα γενικά ε, ήμασταν εξαιρετικά υποστηρικτικοί των χωρών αυτών, με δεδομένο ότι είναι οι μόνες οι οποίες έχουν, είμαστε οι μόνες φορές, ο μόνος οργανισμός που έχει περιφερειακή συμφωνία με τις χώρες αυτές, αλλά είμαστε και επικριτικοί των νέων αυτών κινήσεων, όπου η όλη τάση που διαφαίνεται είναι να κλειστούν οι ανοιχτέ θάλασσες και να ξαναγκαστούν τα σκάφη να λειτουργούν και να λιεύουν μόνο σε πολύ στενότερο βλέπουμε ελάχιστες, να δούμε το χάρτη ουσιαστικά, ελάχιστες θύλακες ανοιχτών θαλασσών. Αυτό το οποίο είναι περισσότερο πρόβλημα είναι ότι η διεθνής ε, ε, διακυβέρνηση που, δίνεται, που, που, που εξασφαλίζεται από το WPFC ε, δεν θα ισχύει από το ενδυτικό δηλαδή Κεντρικό Ειρηνικό δεν θα μπορεί πάρα πολύ να συνεχίσει να δραματίζει το ρόλο του και αυτό θα αντιβαίνει στο οτιδήποτε κάνουμε απανταχού του κόσμου, όπου οι κανόνες οι οποίοι ε, καταρτίζονται από τους περιφερειακούς οργανισμούς εποπτείας δεν ισχύουν μόνο για την ε, ανοιχτή θάλασσα. Στην δυτικό ειρηνικό όμως φαίνεται ότι θα λουσχίσουν τα αντίστοιχα. Extremely worrying, uh, I think, <coughs> is that these countries have introduced a so- το άλλο πρόβλημα είναι ότι οι χώρες αυτές εισάγουν τα λεγόμενα ε, μοντέλα, σχήματα αλλιευτικών ημερών, που είναι ένας ο τρόπος τους πώληση αλλιευτικών δικαιωμάτων. Ε, πουλούν δηλαδή, αν θέλετε, άδειε ε, κατά κάποιο τρόπο, που καθορίζονται σε συνάρτηση με αλλιευτικές ημέρες. Μας ανησυχεί λοιπόν ότι πουλούν όχι μόνο αλλιευτικές ημέρες για την επόμενη αλλιευτική περίοδο, αλλά και για τις μεθεπόμενες. Έτσι λοιπόν οι αλλιευτικές ημέρες ε, έχουν ήδη προποληθεί αρκετά χρόνια πριν, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου καλό για τα αλλιεύματα και τους γόνους όπως φαντάζεστε. Και κάποια τελευταία λόγια σε ό,τι αφορά τον περιφερειακούς κανόνες και την επιστήμη. Η επιστήμη απορράβει από τον WCPFC. Είναι οργανισμός ο οποίος ε, δέχεται τις σχετικές εκθέσεις ό,τι αφορά τα λιεύματα και έχει επιστημονική επιτροπή που μας λέει του πώς κινούνται τα λιεύματα. Περιμένουμε λοιπόν και να έχουμε ανατροφοδότηση ε, σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά θέματα από τον οργανισμό αυτό, γιατί αυτοί παρακολουθούν τα αποθέματα τόνου και δεν θα είχε κανένα νόημα για άλλα αλλιεύματα, αν θέλετε να έχουν τα επικαλυπτόμενα θέματα να έχουν πολύ στενές προσεγγίσεις. Γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό από αμυγός εθνικά όρια, το οποίο ισχύει, αν θέλετε, για τα παράκτια ήδη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αφοσιωμένο, εξειδικευμένο προσωπικό να είναι εγκαταστημένο επιτόπου για την παρακολούθηση εφαρμογή των συμφωνιών, Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι η εφαρμογή των συμφωνιών και η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται σε τοπικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να να έχει κάποια χρηματοδότηση για να στείλει κάποιου συγκεκριμένου προξένου αλληλευτικών πολιτικών κάπου κοντά στην περιοχή ή επιτόπου, προκειμένου να μπορεί το άτομο αυτό να παρακολουθεί άμεσα και ναι, επιστικέπεται τις διάφορες σχετικές χώρες για να εξασφαλίζεται η, εφαρμογή, η σωστή εφαρμογή των συμφωνιών αυτών. Πολύ σωστά επισημαίνεται ότι όντω είναι πολύ απομακρυσμένε οι περιοχέ αυτέ, εξαιρετικά απομακρυσμένε και σίγουρα χρειάζεται να υπάρχουν σχετικοί πρόξενοι αλλιευτικών συμφωνιών εκεί, αλλά βέβαια και πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή των ε, κοινοτικών αντιπροσωπιών εκεί, στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και σε άλλα, άλλα μέρη τη περιοχή. Τώρα, σχετικά με τους παρατηρητές, απευθύνομαι και πάλι στην συνάδελφο να πει κάποια λόγια, που μπορεί να θέλει να αναπτύξει μεγαλύτερη ακρίβεια, αν μου επιτρέπετε. Είναι σύντομο. Πολύ σύντομα. Οι παρατηρητές έχουν υποχρεώσεις στα πλαίσια της Επιτροπής WCPFC και γι' αυτό ε, αυξήθηκαν οι συνεισφορές των πλειοκτητών από 500-1500 ευρώ ε, και είναι υποχρεωτικές. Επιτρέψατε μου κάτι άλλο σχετικά με την περιφερειακή κατάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ ανησυχητική ε, και αυτό έχει επιπτώσεις στην ικανότητα την αλλιευτική. Έχουμε εκεί μια, ένα πολύ μικρό στόλο εκτός από το οικονομικό συμφέρον της αλίας είναι για μας κάποια εγγύηση ότι θα έχουμε κάποια φωνή στην περιφερειακή διακυβέρνηση και ανησυχούμε για την αύξηση της αλλιευτικής ικανότητας κυρίως από τις Ηνωμένε Πολιτείες, η οποία έχει ε, ένα μεγάλο στόλο γρηγρή στην Ταϊουάν, κατ' εξαίρεση των κανόνων των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ε, πλοία με σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να αναφυγούνται στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά υπάρχει, υπάρχουν αυτά τα πλοία, τα μεγάλα πλοία που κατασκευάζονται εκεί εκτός από το σύγχρονο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει αύξηση του στόλου της Ταϊουάν, της Κορέας, της Κίνας και αυτό είναι φαινόμενο ανησυχητικό για την διατήρηση των πόρων, των αλλιευτικών πόρων της περιοχής. Ε, η προσπάθειά μας να συζητηθούν αυτές οι ικανότητες, οι δυνατότητες στην περιφέρεια έχουν πάντοτε απορριφθεί οι προσπάθειές μας, οι προτάσεις μας από τους λεγόμενους συμμάχους, διότι βρίσκουν ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και λεπτό και οι αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκουν ότι είναι άδικο να έχουμε κάτι να πούμε για ε, την, αύξηση των ικανοτήτων. Προτείναμε πολλές φορές ένα πάγωμα, ένα παγκόσμιο πάγωμα ε, των στόλων, των αλλιευτικών ε, αλλίας θηνοειδών. Δεν έχουμε πετύχει κάτι, αλλά είναι ένα σχέδιο το οποίο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη σοβαρά από τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. για να εμβαθύνουμε περισσότερο στο δυτικό ειρηνικό υπάρχει πράγματι αύξηση του δυναμικού. Η ΕΠΑ με ναυλωμένα σκάφη από τον στόλο των Κινέζων και μετά η Κίνα. Η Κίνα αύξησε τα τελευταία δύο χρόνια από 5 πέρασε σε 15 παραγαδιάρικα, σε 12 παραγαδιάρικα διορθώνει η πρόεδρος και έχει και την άδεια να, να κατασκευάσει μέχρι 20 το οποίο είναι μια αύξηση πραγματικά ασύλληπτη, απαράδεκτη. Και επιπλέον η Ιαπωνέζη ε, ζήτησε και ε, ζήτησε την υποστήριξη σε σχέση με το αίτημά τη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει να υποστηρίξει την Ιαπωνία για την αύξηση του δυναμικού όσον αφορά τα παγαδιάρικα και υποστήριξη όσον αφορά την θέσπιση ε, απαγορευμένων ζωνών. Και ξέρουμε ότι έχουν γίνει αυτά τα διαβήματα και ότι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να υποστηριχθεί η Ιαπωνία στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής του Δυτικού Ειρηνικού. Το λέω αυτό και από επαφές με τους Ιαπωνέζους, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε δυνατότητα να το γνωρίζουμε. Και δεύτερον, παρόλα αυτά, καθώς είναι τόσο πλούσια σε αλλιεύματα αυτά τα ύδατα, για το στόκ, τον απολογισμό της κατάστασης, η ίδια η Επιστημονική Επιτροπή ζήτησε μείωση του δυναμικού, μείωση της αλληλευτικής προσπάθειας και το διαβάζω στα αγγλικά του Big Eye, δηλαδή του ξυφοειδούς ε, πατούδο στα ισπανικά, διότι για τον ε, ε λευκόπτερο yellowfin ε, τόνο και για τα άλλα λεύματα είναι σε καλή κατάσταση. Το μόνο το οποίο έχει προβλήματα είναι το ξυφοειδές το Big Eye και γι' αυτό συστήθηκε μια μείωση της αλλιευτικής προσπάθειας, της σύλληψης αλλιευμάτων. Αυτό είναι ένα από, θα έλεγα, τα λίγα σημεία που υπάρχει αύξηση δυναμικού και χώρες ε, όπως η ΕΠΑ που έχουν διαφορετικές θέσεις όσον αφορά το θέμα της μείωσης ε, ε, της αλληλευτικής προσπάθειας και της αηφόρου ανάπτυξης είναι ένα συμβαλόμενο μέρος στο δυτικό ειρηνικό που έχει αυξήσει την αλληλευτική προσπάθεια εκεί. Αυτό συμβαίνει στην καθημερινή πραγματική ζωή. Ο, κάποιοι κάνουν ό,τι τους ε, γουστάρει, αλλά αυτή είναι η ζωή στην Αλία και ε, αυτό είναι ενδιαφέρον. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώθηκε το σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη. Όχι, όχι, εντάξει. Χρονοδιάγραμμα λέτε. Μάλιστα, χρονοδιάγραμμα είναι κάπως πιεστικό το χρονοδιάγραμμα. Παρουσίαση 25-26 Ιανουαρίου 2011, 15-16 στη συνέχεια ψηφοφορία και ε, παρουσίαση στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να ε, μπορέσουμε τα, τα του δυτικού ειρηνικού, κεντρικού ειρηνικού να έχουμε πληροφορίες. Θα προσπαθήσω να έχω τις πληροφορίες στην έκθεση μέχρι αυτή την ημερομηνία και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα το οποίο να αξίζει να ενταχθεί στην έκθεση αυτή που είναι υπό ε, σχεδιασμό θα σας ζητούσα να αναβληθεί το χρονοδιάγραμμα αυτό για αυτό το θέμα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το σημείο 9. Αύριο θα συνέλθουμε πάλι στις 9 θα συναντηθούμε. Τώρα έχουμε συνάντηση συντονιστών. Σας ευχαριστώ. Α, συγγνώμη. Με ενημέρωσαν αποστεριόρι ε, με ε, ε καθυστέρηση ότι θα είναι η τελευταία λέει συνεδρίαση αυτή διότι... Α, ότι εσείς αποχωρείτε λέει. Σωστά, συνταξιοδοτήστε. Μάλιστα, έχετε την τύχη να πάτε σε συνταξιοδότηση. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Φιλοδοξία κάθε υπαλλήλου να φτάσει στην ηλικία συνταξιοδότησης. Και εγώ το έχω καθαρά υπόψη αυτό, ναι. Εν πάση περιπτώσει, διαβιβάστε, διαβιβάστε παρότι θα προσπαθήσω να τηλεφωνήσω συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες από αυτή την Επιτροπή για την καλή συνεργασία που πάντα είχαμε με ένα υποδειγματικό υπάλληλο που ήταν ο κύριος Σόκουες. Το λέγω αυτό ειλικρινά. Ευχαριστώ.